Okay, colleagues, we're giving everybody the obligatory minutes on a Monday. Συνάδελφοι, έχουμε δώσει σε όλους το ακαδημαϊκό τέταρτο για να έρθουν ε, εδώ Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσία σας εδώ. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη ή έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν ε, έχω αιτήματα για αλλαγή. Μπορούμε να την εγκρίνουμε όσο έχει. Ωραία, ευχαριστώ. Σημείο 2 Ανακοινώσει της Προέδρου. Την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο θα γίνει μια κοινή ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Υποεπιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους νικητές του βραβείου Ζαχάροφ ε, οι αντουφρονούντες στη Βενεζουέλα πέραν το βραβείο. Η συνεδρίαση θα γίνει παρουσία της ε, ε Ευρω, ε, της Eurolat, της Eurolat και θα γίνει από τις 7.30 μέχρι τις 9 στην αίθουσα νη ΝΙΕΝΑ4. Φαντάζομαι θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για αυτή τη συνεδρίωση. Αυτά λοιπόν για το Στρασβούργο και μία ακόμα ανακοίνωση. Δεν υπάρχει διερμηνία από τα πολωνικά σήμερα. Δεν βλέπω βέβαια συναδέλφους ε, Πολωνούς εδώ σήμερα. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Λέντα που ε, είναι γλωσσομαθής ε, θα τα καταφέρει. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων τις 23 Σεπτεμβρίου έχετε τα πρακτικά. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αλλιώς θα θεωρηθούμε ότι εγκρίνονται. Σημείο 4. Έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών. Έχετε τα πρακτικά τη συνεδρια 21 21η Νοεμβρίου και πάλι για τυχόν παρατηρήσει, ε, διαβιβάστε στη γραμματεία μέχρι το τέλο τη συνεδρίασης. Αν δεν ε, λάβουμε παρατηρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα ή μάλλον θέματα. Θα συζητήσουμε τα θέματα 5 και 6 μαζί. Απαλλαγή ε, του Γενικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και αναθεώρηση για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ε, περί τίνος πρόκειται, για εκείνους που δεν γνωρίζουν την απαλλαγή και για τους προσκεκλημένους μας εδώ σήμερα. Η απαλλαγή είναι μια διαδικασία βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο πώς ε, εκτελέστηκε ο προπολογισμό και ε, εξετάζουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζουμε τις γραμμές προπολογισμού ε, της αναπτυξιακής στο βασικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο όπως ξέρετε είναι εκτός προπολογισμού της Ένωσης και βασίζουμε το έργο μας στην ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Γνωμοδοτούμε λοιπόν για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Η συγητή ε, για τι γνωμοδοτήσει, συντάκτη μάλλον, είναι ο κύριο Φρουντσούλικα, ο οποίο απουσιάζει σήμερα. Ο Ρόμπερτ Νόιζερ είναι αυτό ο οποίο ε, θα ε, παρουσιάσει εκ μέρου του. Νόρμπερτ Νόιζερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ο συντάκτη τη γνωμοδότηση μου ζήτησε να λάβω το λόγο εξ του. Επαναλαμβάνω ότι ε, παρά το γεγονός ότι ε, υποστηρίζουμε τη χρήση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης ε, για κάθε περίπτωση και για να δώσουμε και νέα όθηση σε μηχανισμούς ελέγχου που εξετάζουν ε, την ε, ε, κατάσταση των χωρών αποδεκτών των πόρων κατά της διαφθοράς και εκφράζεται ανασυχία για τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση ε, κινητοποίηση των ταμείων σε συμβάσει ελέγχου του προπολογισμού. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, αυξήσει την ε, ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση προ τι χώρε εταίρου για τι δυνατότητε χρηματοδότηση και να διευκολύνει τη χρήση του. Επίση, όπω αναφέρεται στη γνωμοδότηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό η το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται και να τη χάνει διαβούλευση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του 11ου ε, αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο υποτίθεται ότι θα λάβει υπόψη του και το θεματολόγιο για το 2020 και τη νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ανάπτυξη, ε, σεβόμενη και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης. Τέλος, ε, προσδίδω ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός κλάδος εάν συμμετέχει για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πράγματι, ο δημόσιος τομέας από μόνος του δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για επενδυτικά προγράμματα δημοσίου συμφέροντος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορεί να είναι χρήσιμο να υπάρξει μια ε, σύμπραξη, να χρησιμοποιείται το blending, ε, να υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί διαφάνειας ε, και να εφαρμόζονται αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφο το λόγο για την απαλλαγή η Χάιντι Χάουταλα και ο κύριος Σαφχάζερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ το σχέδιο γνωμοδότησης του κύριου Φρουντζούλικα. Χαίρομαι που τονίζει το ρόλο των Ευρωπαϊκών Πιστητικών Οργανισμών και υπάρχει κατάλληλη αναφορά σε αυτά στη γνωμοδότησή του. Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι λυπούμαστε πολύ που οι αρχές της αποτελεσματικής ανάπτυξης φαίνεται να οδηγούν σε βραχυπρόθεσμα συμφέροντα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώνουμε ότι δεν είμαι μόνο εγώ ή εμείς που μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αναφέρεται και στην ενδιάμωση ε, αξιολόγηση και του DCI και του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου του Μηχανισμού για την ε, Συνεργασία για την Ανάπτυξη. Ε, και το βασικό παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι ε, το μέσο που συνεισφέρει στη σταθερότητα και την ειρήνη, που αμφισβητείται ως προς το νομικό του σκέλος. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το όλο ζήτημα της δαπάνης κονδυλίων για την επανένταξη όσων επιστρέφουν στο Αφγανιστάν. Το ελεγκτικό συνέδριο έκανε πάρα πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις για την πολιτική για τα βιοκαύσιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαιτεί εθελοντικά προγράμματα για να επαληθεύσει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων που εγκρίνει ε, δεν ε, δημιουργεί πολύ σημαντικούς κινδύνους ε, για το περιβάλλον και την κοινωνία, για παράδειγμα καταναγκαστική εργασία παιδιών, φτωχές συνθήκες εργασίας ε, και θέματα ασφάλειας και προστασίας. Και υπάρχει και η νομοθεσία iLook τη αλλαγή τη χρήση γεών για την βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων. Δεν καλύπτεται αυτή από την αξιολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να είμαστε αρκετά αυστηροί επ' αυτού, διότι ε, ακολουθούμε μία οδό που δεν είναι καλή για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους φτωχού ανθρώπους που ζουν εκεί. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα στους κανόνες διεξαγωγής των μειοδετικών διαγωνισμών και προμήθειες και αυτό είναι συνεχές πρόβλημα και κάθε φορά το ελεγκτικό συνέδριο θίγει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ε, Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, γιατί οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου δεν έχουν, τόσες πολλές, έχουν τόσα πολλά σφάλματα σε σχέση με τον DCI. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και επίσης ε, χαίρομαι για τα συμπεράσματα του ε, ελεγκτικού Συνεδρίου ε, για το γεγονός ότι η δαπάνη για τι εξωτερικές δράσεις είναι αυτή η οποία περιλαμβάνει τα λιγότερα σφάλματα. Είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε ε, περήφανοι δεδομένων και των δύσκολων συνθήκων των οποίων δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ισηγητά για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά την εκτέλεση του 2016 για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Όμως κάποια στοιχεία θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τονιστούν περισσότερο. Δεν διαφωνώ με την αρχή της προσφυγής ε, της υποστήριξης από τον προπολογισμό για την εκτέλεση του Ταμείου Ανάπτυξης, όμως συμφωνώ με τις ανησυχίες του εισηγητή σε σχέση με την καταλληλότητα της αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Αναπτυξιακής Βοήθειας, ειδικότερα για τις χώρες της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να ορίσει με ε, πιο σαφή και πιο ακριβή τρόπο τους στόχους αυτής της αναπτυξιακής βοήθειας και των προγραμμάτων, όπως επίσης και σημαντικές εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αρκούν ε, στο να ε, μπαίνουν σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο εκατομμύρια ευρώ κάθε ε, χρόνο. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ε, να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε τη χρήση αυτών των κονδυλίων σε σχέση με το σεβασμό των μειονοτήτων και την πραγματική ανάπτυξη. Επομένως, ε, όλα αυτά που περιλαμβάνει η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου θα έπρεπε να μας ανησυχήσει γιατί λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν αρκετά ε, ακριβής όσον αφορά τις προηγούμενες αξιολογήσεις της, ούτε λαμβάνει υπόψη κατευθυντήριες γραμμές. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχω πραγματικά πάρα πολλές αμφιβολίες ε, σε σχέση με την μεικτή προχρηματοδότηση ιδιωτική και δημόσια του προγράμματος αυτού. Αν ισχύει το γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με το 11ο Ταμείο ανάπτυξης ε, με 30,6 δις ευρώ δεν μου φαίνεται ε, αυτή η νικτή χρηματοδότηση ο καλύτερος τρόπος. Ο κίνδυνος είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα να επικεντρωθεί περισσότερο σε τμήματα συγκεκριμένα των οικονομιών των χωρών αντί σε υποδομές που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον πληθυσμό όπως τα νοσοκομεία, τα λιμάνια, οι αγορές, οι δρόμοι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο για τη δουλειά ε, των για την ζωή των ανθρώπων αυτών και αυτά μπορούν να προέλθουν μόνο από δημόσιες δαπάνες. Επίσης το θέμα της, του δημόσιου συμφέροντος. Όλα αυτά πρέπει να προκύπτουν, να έχουν ένα αποτέλεσμα για τους πολίτες των χωρών αυτών. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη σοβαρά το γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση αποκλίνοντα ιδιωτικά συμφέροντα να δημιουργούν προβλήματα για μια επικίνδυνη κατάσταση στι χώρες αυτές και μπορούν να θέσουν και ένα αμφιβόλο την ανεξαρτησία και την κυριαρχία στοιχεία των κρατών ε, στα οποία θα υλοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σαφχάουζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τώρα μόλις γύρισα από την Κεντρική Αφρική, πάω κάθε μήνα, όπως είναι και ο προγραμματισμός μου, φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που είχα ε, και εγώ ε, καταλήξει ε, μόλις βγήκα από το αεροπλάνο την Κυριακή το πρωί. Όσον αφορά το Ταμείο του Μπεκού και ε, αυτό που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα με την δημιουργία ενός ε, ταμείου, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστό. 25 και πάνω χρόνια εμπειρία έχω, 30 χρόνια, για να μην σα κρύβω και την ηλικία μου, 30 χρόνια ε, με, ενασχόλησης με την αναπτυξιακή πολιτική στην Αφρική. Ο εισηγητή τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό. Αυτό εγώ ε, συγκρατώ και έχω παρατηρήσεις να κάνω σε σχέση με τον Διευθυντή ε, για τα ζητήματα ανάπτυξης, ε, γιατί η Κεντροαφρική αφρικανικές χώρες θα ήταν σε θέση να λειτουργήσουν μέσω αυτού του ταμείου ή όπως έχει γίνει άλλες φορές μια πλατφόρμα να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών όπου όλοι οι δωρητές και τα αρμόδια υπουργεία, οι εμπλεκόμενοι φορεί ε, που ενδιαφέρονται, για παράδειγμα οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, να μπορούν να συντονιστούν για να επιτύχουν του στόχου. Αυτό είναι ουσιαστική σημασία αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Άρα, ε, νομίζω ότι το σημείο 2 είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα, σημείο 4, πάρα πολύ καλό και αυτό. Δεν πρέπει να συγχέουμε τα, τα ιδιωτικά και τα ε, δημόσια κονδύλια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλω, ας πούμε, να έρθω με μια επιχείρηση που είναι ηγετική στον τομέα της ε, γεωργίας και του κρέατος, για παράδειγμα. Ε, το πρώτο πράγμα που μου λέει η επιχείρηση είναι δεν έρχομαι γιατί δεν έχω ασφάλεια. Πώς θέλετε λοιπόν να υπάρχει ε, επένδυση και ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Δεύτερον, αν θέλετε να κάνετε ένα σφαγείο για παράδειγμα, χρειάζεται ηλεκτρισμό χρειάζεστε δρόμους, χρειάζεται ένα σύστημα ψήξης. Ε, τώρα φανταστείτε το κρέας, το σκοτώνουμε, το σφαγιάζουμε με κάτι χιλιάδες μύγες που πέφτουν πάνω και μετά στη συνέχεια μεταφέρεται. Εγώ παίρνω αντιβίωση γιατί πλέον ε, το κύκλωμα της ψήξης δεν λειτουργεί πια στην, ε, ανάπτυξη, στην Αφρική. Δεν υπάρχει πλέον ψήξη για τα προϊόντα κρέατος. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, χρειάζεται μια ιδιωτική επένδυση, η οποία θα γίνει, αλλά πρέπει να συνοδεύεται αυτή η επένδυση από μια δημόσια επένδυση. Συνεπώς, η σημασία ενό συντονισμού, χωρίς να τα συγχαίουμε μεταξύ τους, πρέπει να υπάρχει όμως πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο. Αν θέλετε να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη, το ίδιο πρόβλημα έχετε να αντιμετωπίζετε. Αν κάποιος, για παράδειγμα, θέλουμε να έχουμε ε, μελισσοκομεία, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ε, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ε, τους γεωργούς, σε όλη τους την προσπάθεια. Χρειάζονται βασικά στοιχεία. Ή ας πούμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πτυνοτροφείο, πρέπει να υπάρχει το ε, τα, τα απαραίτητα ώστε να τραφούν ε, τα κοτόπουλα. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, ότι πρέπει ε, η ιδιωτική επένδυση να συνδυαστεί σε μια βασική, με μια βασική δημόσια επένδυση. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να το, να το πετύχουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Κεντρική Αφρική και το βλέπω αυτό σήμερα, ε, είναι πάρα πολύ πιθανό κατά τα τελευταία χρόνια ε, έχουν υπάρξει σχετικές εκτιμήσεις. Το Καμερούν, ε, το Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, ξέρετε την κατάσταση, το Σουδάν, όλη αυτή η κεντροαφρικανική περιοχή, το γνωρίζετε πολύ καλά τίποτε τελικά δεν θα πετύχουμε με, με το βόρειο τμήμα της Αφρικής που γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν η, η Αλγερία, η Λιβύη, η Αίγυπτος ε, αν και η Κεντρική Αφρική εκραγεί με όλες αυτές τις ε, ε, χώρες, που, κυρίως αυτές που γειτονεύουν με το βόρειο τμήμα, θα είναι η κατάσταση δραματική η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει καθοριστική σημασία ε, συμμετοχή με τη βοήθειά της και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, το Φεβρουάριο θα ξαναπάμε εμεί με την αποστολή μα. Ε, θα πάτε κι εσεί και ο Κριστιανό θα πάει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και πολύ χρήσιμο θα είναι το υπόβαθρό σα, η εμπειρία σα, ε, ο προγραμματισμό ε, τη προσπάθειά μα, βοήθειά μα πρέπει να είναι αυτό που είπατε κι εσεί. Πρέπει να δώσουμε τι προτεραιότητε, αλλά κάθε, κάθε χώρα πρέπει να έχει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα, να πρέπει να παντρευτεί ο ιδιωτικό με το δημόσιο τομέα με τον τρόπο που αναφέρατε. Ο Σαλ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ερώτημά μου ε, όσον αφορά το πρώτο σημείο και τη βοήθεια από τον προπολογισμό, το πρώτη, πρώτο σημείο που δεν είναι εδώ εισηγητή βέβαια, αλλά μπορεί να, μας, να μου απαντήσει ο κύριο Νόιζερ ενδεχομένω. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν είναι και εδώ κάποιο από το ελεγκτικό συνέδριο. Όχι. Τουλάχιστον κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω να μου απαντήσει. Εγώ να καταλάβω καταρχά κάποια πράγματα. Ποια ήταν η μέθοδο που εφαρμόστηκε για να καταλήξουμε στα ε, συμπεράσματα αυτά και ε, στα σχέδια σύμφωνα με τα οποία ε, η βοήθεια αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Προφανώ μπορεί να βελτιωθεί, αλλά τι ακριβώ μέθοδος ακολουθήθηκε. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε κάποιο έγγραφο, που πούμε, το οποίο υποβλήθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο από τις ε, ε, αρχές ε, τις υπεύθυνες για τον προϋπολογισμό των χωρών τις οποίες εξέτασε οι χώρες δικαιούχοι, αποδέκτες της βοήθειας έχουν μια επιτροπή προπολογισμού σε ένα κοινοβούλιο που δουλεύει ορθά ή τα αποτελέσματα ας πούμε ε, είναι καλύτερα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει μια σωστή επιτροπή προπολογισμού σε σχέση με άλλες. Υπάρχει λοιπόν μια αποστολή, μια, συγγνώμη, επιτροπή ε, ε και ελέγχου αυτών ε, του προπολογισμού. Θα ήθελα να τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα και θα ήθελα επίσης να ξέρω τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτόν τον έλεγχο. Και κάνω αυτές τις παρατηρήσεις γιατί πριν από μερικά χρόνια εδώ στην Επιτροπή μας ε, υπήρχε μια έκθεση του κύριου Πίνγκστον που ήταν μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και ο οποίος ε, είχε εκφράσει κάποιες επικρίσεις ε, σε σχέση με κάποιες αφρικανικές χώρες και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του προϋπολογισμού και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και είχε πει ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική η κατάσταση ε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αφιερωθεί στο σκοπό αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι πλέον έχουν μειωθεί γιατί πρέπει να γίνονται περικοπέ στους ανθρώπινους πόρους παντού πλέον και από την άλλη θέλουμε ένα μέγιστο αποτελεσματικότητα. Ε, θα γίνει αυτό. Ε, θα θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότεροι να ασχολούνται με, τον, ε, με, τα θέματα ε, της αναπτυξιακής βοήθειας και της, του, ε, της βοήθειας και του, της εκτέλεσης του προπολογισμού. Από την άλλη θέλουμε περικοπές και μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ε, πώς θα γίνουν και τα τρία μαζί. Αυτές είναι λοιπόν τεχνικές ερωτήσεις, οι οποίες όμως έχουν σημαντικές πολιτικές συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να, πάρει, να θέλει να πάρει το λόγο. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπαγκιούρα από την ΤΕΦΚΟ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσετε κάποια από τα ερωτήματα του κυρίου Γκέρεντς, για παράδειγμα, τα πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να επανέλθω σε μερικά ζητήματα, είτε ερωτήσεις είτε στοιχεία τα οποία έθεσε ο εισηγητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για ε, την ε, ε, συμμετοχή τους στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμών. Εμείς ε, εκτιμούμε την υποστήριξη της Επιτροπής σας ε, στην δημοσιονομική υποστήριξη. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει τέλος πάντων κάποια σταθερότητα στην ανάμιξη, στο μείγμα των ε, προγραμμάτων του χαρτοφυλακίου της αναπτυξιακής μας συνεργασίας. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τις τρίτες χώρες να σας πω το εξή ότι από τη σημαντική μεταρρύθμιση του 2011 υπήρξε μία ανακοίνωση που στόχευε την αναθεώρηση της δημοσιονομικής υποστήριξης, κάναμε αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών κάτω, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαίου δικαιώματα, όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα προγράμματα δημοσιονομικής υποστήριξης βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Ε, το ίδιο ισχύει για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Στο παρελθόν ε, υπήρξαν κάποια, κάποιες ομάδες παρακολούθησης οι οποίοι την ασχοληθεί ειδικότερα ε, με τα προγράμματα αυτά και μετά από, την παρατήρηση, τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου κάναμε και ε, ε, στις, όσον αφορά τις Ονδούρες μια πολύ, σημαντική προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης. Μπορώ να σας δώσω και τα αριθμητικά στοιχεία αν θέλετε που αφορούν την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών είτε εκεί είτε σε αντιπροσωπείες. Ε, όσον αφορά τώρα την έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου, πρέπει να πω ότι είναι μάλλον θετική όσον αφορά την ε, ενεργοποίηση των ε, εγχωρίων πόρων, ε, ουσιαστικά η δημοσιονομική υποστήριξη μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική. Οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου είναι χρήσιμες και έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις νέες κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε δημοσιεύσει και έχουν συζητηθεί με το ελεκτικό συνέδριο το Νοέμβριο του 2017. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη σοβαρά και την έκθεση και τις ε, συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Όσον αφορά τώρα την, τον ΠΕΚΟΥ και ε, προφανώς τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Ε, ναι, η συνεργασία και ο συντονισμός των δωρητών είναι ένα καταλυστικό στοιχείο, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το καταπίστευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιφέρει τη θέμενη αξία. Και το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του το αναφέρει. Πρέπει βέβαια να βελτιωθεί περαιτέρω ο συντονισμός. θα υπάρχει καλό συντονισμό αν γίνει γύρω από την κυβέρνηση. Ε, για παράδειγμα, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ε, Δημιουργίας Ειρήνης ε, είναι το πρόγραμμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την ηγεσία όπως επίσης και τη συνεργασία με την κυβέρνηση της ε, Κεντρικής Αφρικής. Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω για τα στοιχεία συγκεκριμένα που αναφέρει ο εισηγητής στην έκθεσή του. Ίσως εμείς ε, να ερμηνεύουμε πιο θετικά ε, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ποτέ έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που διάβασα τόσο θετική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό λέω ότι είναι σχετικώς θετική για το καταπίστευμα Μπεκού που είναι κάτι το ε, πολύ ε, σημαντικό και είναι κάτι το περίπλοκο προκειμένου να υλοποιηθεί. βεβαίω, ε, οι συστάσεις ε, θα συμπεριληφθούν στις νέες κατευθυντήριες ε, γραμμές, οι οποίες βεβαίω αναθεωρούνται αυτή τη στιγμή και θα δημοσιευθούν Οκτώβριο του 2018 και επίσης θα επεξεργαστούμε ένα αίτημα του ελεγκτικού συνεδρίου περισσότερο που είναι μια λεπτομερέστερη περιγραφή των κριτηρίων που ε, δίνουν τη δυνατότητα εκ των προτέρων ε, να ε, δούμε την προστιθέμενη αξία του κάθε καταπιστεύματος που θα δημιουργείται στο, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού το είχαμε κάνει αυτό, κατόπιν ε, σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προηγούμενη απαλλαγή. Για σκοπό είχαμε να βελτιώσουμε την ορατότητα των προγραμμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, γνωρίζοντας βέβαια ότι μπορούσαμε περισσότερο να περάσουμε μέσω του συστήματος του ΟΗΕ ή της Παγκόσμιας Τράπεζας και θα μπορούσαμε να το κάνουμε ευκολότερα έτσι και μέσω της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ένα ακόμη σημείο που μου φαίνεται σημαντικό στο πλαίσιο πλαίσιο της έκθεσης ε, που αφορά την αναθεώρηση, την, ε, την μεσοπρόθεσμη ε, την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αναθεώρησης αυτής, γιατί η νομική βάση και μιλάω για το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ταμείου ε, αναπτυξιακής ε, ε, συνεργασίας. Θα σας ενημερώσουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, μέχρι το τέλος χρονιάς δηλαδή, θα έχετε την έκθεση στα χέρια σας. Η αναθεώρηση αυτή ε, ούτως ή άλλως γίνεται στο πλαίσιο της, πολιετούς, του πολιετούς προγραμματισμού. Ο Στέφανο Μαρσεβίση θα είναι εδώ για να σας τα πει πιο μετά. Ε, και πιστεύουμε ότι βέβαια έτσι θα έχουμε μια καλύτερη σχέση και με την επίτευξη, με, με την, ε, μια καλύτερη σχέση με το πώς πάει η ε, επίτευξη των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά τώρα του μειοδοτικού διαγωνισμούς ε, και αυτό που με ρωτήσατε, γιατί εμείς, εμείς ε, έχουμε ε, το ίδιο περιβάλλον ελέγχου και για το Ταμείο ανάπτυξη, που αφορά περισσότερο τις χώρες ΑΚΕ, ενώ για τις για το, για το μέσο αναπτυξιακή συνεργασίας είμαστε περισσότερο στην Ασία ε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην Ασία. Όντως υπάρχουν κάποια σφάλματα, αλλά τα σφάλματα προέρχονται από την έλλειψη εγγράφων. Δεν είναι ότι υπήρχαν ατασταλίες, δεν μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι δεν υπήρξαν ατασταλίες, γιατί δεν υπήρχαν όλα τα έγγραφα στη διάθεσή μας. Το ε, ποσοστό υπολοιπωμένου σφάλματος είναι 1,67%. Ένα ποσοστό το οποίο βρίσκω ότι είναι ε, αρκετά εξαιρετικό σε ένα περιβάλλον εφαρμογής πάρα πολύ περίπλοκο. Βεβαίως ε, θα ε, εξετάσω πιο προσεκτικά αυτό το οποίο αναφέρατε και όσον αφορά το θέμα των, της σύναψης συμβάσεων για τις προμήθειες, ναι, ευχαρίστως να επανέλθω για, με, τα συμπεράσματά μου. Σάρλο, σου απαντά αυτό την ερώτησή σου. Ναι, ναι, έχω μια ερώτηση για τον πρακτικό τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. Έχετε αντιπροσωπείες ε, στις χώρες ε, που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση, υπάρχουν ε, υπεύθυνοι που παρακολουθούν πιο στενά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια από τον προϋπολογισμό. Υπάρχει κάποιος στην κεντρική διοίκηση ή τουλάχιστον κάποιος στο τμήμα προϋπολογισμού ε, το οποίο εξετάζει αυτές τις διαφορές ή έγιναν μόνο κάποιοι εκ των υστέρων έλεγχοι. Καταρχάς, ε, το προγράμματα αυτά του προπολογισμού είναι προγράμματα τα οποία τα παρακολουθούμε κεντρικά. Ε, δεν υπάρχει κάποιος επιτόπου, υπάρχουν κάποιοι για τον πολιτικό διάλογο με τους εταίρους, για την παρακολούθηση των δικτών επίσης ε, που ε, μπορούν να οδηγήσουν και στην εκταμίεση των διαφόρων δόσεων. Αλλά η, τα στοιχεία, τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, εξετάζονται πάντα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου το, το οποίο εξετάζει τα θέματα αυτά. Και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ή κάποιε αμφιβολίε, μπορούμε να τα παραπέμψουμε σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο επιτρόπου, για να δούμε τι συνθήκε τη χώρα πριν ξεκινήσει μια ε, διαδικασία υποστήριξη στον προπολογισμό από εκεί και πέρα ε, γίνεται ε, έλεγχος ε, πριν ε, δοθεί μια θεώρηση για την διαδικασία και από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες πριν, γίνει, πριν δοθεί αυτή η έγκριση ελέγχουν την κατάσταση. Αν είναι σύνθετα τα πράγματα, πάλι περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο ε, προεδρεύει ο Γενικό Διευθυντή. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τι αντιπροσωπείε βεβαίω ε, ε, επιτόπου μόνε του. Υπάρχει πάντα κάποιο εκπρόσωπο, αλλά καθημερινά υπάρχουν ομάδε επιτόπου, οι οποίε παρακολουθούν την υποστήριξη στον προπολογισμό και όπω σα είπα, δεν είμαι τώρα σε θέση να σας πω ποιοι είναι αρμόδιοι ποιο είναι ο αριθμό αυτών των ανθρώπων. Τελευταία ερώτηση. Τι ρόλο έχουν λοιπόν οι εθνικέ αντιπροσωπείε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο αποκαλείται εθνικέ αντιπροσωπείε είναι οι εταίροι, οι κυβερνήσει δηλαδή, οι αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στις χώρες που βοηθούμε. Α, ο ρόλος της αντιπροσωπείας είναι καταρχάς να γίνεται αυτός ο καθημερινός διάλογος ε, με ένα τεχνικό κλιμάκιο το οποίο μπορεί να λάβει τα χρήματα, διότι τα χρήματα ορισμένες φορές εντάσσονται στον προπολογισμό είτε για κάποιο κλαδικό πρόγραμμα, ή τον τομέα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν διάλογος ε, για την εξέταση της κατάστασης, για τους στόχους τους οποίους πρέπει να επιτύχουμε Στη συνέχεια, όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι, η αντιπροσωπεία συντάσσει για πρώτη φορά το φάκελο για να είναι βέβαιοι ότι ε, μπορούν να κάνουν την αίτηση για τις πληρωμές. Αλλά η αντιπροσωπεία είναι επί τόπου, πολύ κοντά στις εθνικές αρχές για να δει τα θέματα τα οποία είναι αρκετά περίπλοκα να βοηθήσει για να υπάρχει λοιπόν και μια δεύτερη αξιολόγηση στη συνέχεια που γίνεται επί τόπου και να δοθεί μια δεύτερη σύνταξη φακέλου. Μία ακόμα ερώτηση γιατί περιμένει και ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Σαφχάουζερ. Τελευταία ερώτηση. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια εμπειρία για όλες αυτές τις τυπικότητες. Όλη αυτή οι τοπικοί, ε, ε τυπικοί μπορεί να παρουσιάζονται σε οτιδήποτε. Παραδείγματος χάρη, πρόσκληση ε, προκήρυξη διαγωνισμού. Μιλάω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ε, κατακυρώνονται σε μια κινέζικη εταιρεία. Έξι μήνες μετά λοιπόν φαίνεται ότι μπορούν να γίνουν. Ε, να μην εμπιστευόμαστε λοιπόν τα όσα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για τον προπολογισμό, γιατί, για το διαγωνισμό, γιατί πολύ συχνά είναι ε, παραπλανητικά τα στοιχεία και πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά. Διότι μπορεί να κρύβεται και ε, ε, επεξαίρεση κονδυλίων και να υπάρχουν προβλήματα. Είναι πολύ εύκολο να γνωρίζουμε. Ξέρουμε, για παράδειγμα, πόσο στοιχίζει η κατασκευή ενό χιλιόμετρου δρόμου, η ανακαίνιση ενό νοσοκομείου. Όσοι έχουν εμπειρία με ανάπτυξη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και βλέπουν κατά πόσον υπάρχουν ατασταλίε. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, για παράδειγμα. Σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια καταστροφική κατάσταση, θελήσαμε να αγοράσουμε για πολλά εκατομμύρια ε, ε, ευρώ. Η γεωργία δεν αρκεί ούτε καν για να ζήσει ο πληθυσμό στη χώρα και θελούσαμε να αγοράσουμε. Δεν είχε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση, ήταν από άλλη χώρα. Ε, εξοπλισμό, μηχανικό. δεν μπορούν ούτε να επισκευάσουν τα οχήματα. Επομένως πρέπει να αγοραστεί, αγοράζεται ο εξοπλισμό, αλλά μπορεί να μην υπάρχουν δρόμοι, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να μάθουν πώς να οδηγούν αυτά τα οχήματα και είναι καταστροφή. Και γιατί δίνονται όλα αυτά τα κονδύλια, διότι επιτρέπουν να διαρρεύσουν στη συνέχεια στα διάφορα δίκτυα. Ε, αυτά λοιπόν για να τα γνωρίζετε και όλα αυτά πίσω από τη στήριξη στον προπολογισμό. Ε, βέβαια η συζήτηση εδώ είναι για την απαλλαγή. Ξέρω ότι η αντιπροσωπεία πρέπει να κάνει αξιολόγηση για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ένα τελευταίο σχόλιο από την Κομισιόν. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία τίθενται. Δε, δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα για τη Γενική Διεύθυνση. Αύκο τίποτα το συγκεκριμένο. Ε, ως εκ τούτου πάμε πίσω στον κύριο Νόιζερ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, Νόρμπερτ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να προσπαθήσω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αφενός ε, θα πρέπει να έχουμε ε, κατά νου ότι ένα κράτος για να πάρει βοήθεια από τον προπολογισμό θα πρέπει πρώτα να είναι επιλέξιμο. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Γιατί κάπως δημιουργείται η εντύπωση ότι όλα τα κράτη μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό. Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να καλύπτουν κάποια κριτήρια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στον ε, προϋπολογισμό είναι πολύ βασικό να υπάρχουν ε, στόχοι. Οι στόχοι λοιπόν που έχουν σχέση με την βοήθεια από τον προπολογισμό ε, θα πρέπει οι στόχοι αυτοί που ετέθησαν το 2011 ε, να αναφέρονται και στους ε, στόχους του προπολογισμού. Σχετικά με την Κεντρική Αφρική, πράγματι νομίζω το Φεβρουάριο ε, θα μεταβεί ε, μια αντιπροσωπεία στην ε, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής. Και όταν πρόκειται για τον συντονισμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, προφανώς και όλοι είναι υπέρ αυτού. Αλλά θα πρέπει να μιλάμε και να ξέρουμε και για τα πότε μπορούμε να μιλάμε για καλό συντονισμό. Η τελευταία παρατήρηση αφορά τα προβλήματα στα οποία εκτίθενται οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως και αντιπροσωπείες οποίες ακολουθούν ε, συγκεκριμένες εντολές. Όμως ε, ο ρόλος ε, που πρέπει να καλύπτει επιτόπου οι κανόνες διπλωματικοί που πρέπει να τηρούνται, αυτό νομίζω είναι λιγάκι δύσκολο και από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι οι αντιπροσωπείες είναι πολύ αυστηρές, μερικές φορές ε, καταργούν κάποια προγράμματα και λένε ότι ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι καλύπτονται κάποια κριτήρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει και την ανάλογη εντύπωση στις ε, άμεσα ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις. Κάθε Σεπτέμβρη έρχονται εδώ οι πρέσβεις των αντιπροσωπιών ε, και συναντιόνται στο Κοινοβούλιο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Μερικές φορές ρωτάμε πώς τα καταφέρνουν ε, επί τόπου. Ε, ίσως μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό, το Σεπτέμβρη που θα έρθουν, ε, να το ξανακάνουμε. Πολύ ωραία. Επόμενη λοιπόν... Ε, τρίτη θα ε, ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό και μετά θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7. Βλέπετε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΕΔΕΦΚΟ, ο κύριος Στέφανο Μανσερβίση, είναι παρόν. Εκεί θα μιλήσουμε για την ενδιάμεση επανεξέταση του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Νομίζω θα μιλήσετε περισσότερο για το έγγραφο προγραμματισμού, γιατί συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, σχετικά ε, με τα εργαλεία της ε, ενδιάμεσης επανεξέτασης. Ε, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουν οι συνάδελφοι ποιε είναι οι διάφορε φάσει που προβλέπονται. Γιατί γίνονται πάρα πολλέ ε, συζητήσει στο Κοινοβούλιο σχετικά με την μακροπρόθεσμη προοπτική του πολιτού σε δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, νομίζω ότι είναι καλό να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι αγαπητοί συνάδελφοι, η ενδιάμεση επανεξέταση του προγραμματισμού, εκεί ακριβώς έχουμε το δικαίωμα του ελέγχου. Και νομίζω αυτό θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο, κάπου στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτή λοιπόν είναι και η δική σας ευκαιρία να ε, κάνετε ερωτήσεις για τον προγραμματισμό. Το θέμα που τίθεται είναι ε, δαπανάμε τα χρήματα όπως ακριβώς ε, προβλέπετε ή όχι. Αυτή τη συζήτηση κάναμε πριν έρθετε και σχετικά με την απαλλαγή. Κύριε Γενική Διευθυντά, παρακαλώ έχετε το λόγο. Νομίζω ότι ευχαριστώ πολύ Λίντα. Όπως ε, ακριβώς ε, προβλέπετε, κυρίως ε, όσον αφορά την προγραμματική περίοδο, αυτό που εξετάζουμε είναι τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με την εφαρμογή των προγραμμάτων για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο οι διάφορες χώρες ακολουθούν ε, τις ε, προτεραιότητες όπως πρέπει και επίσης εξετάζουν και το θέμα του διαλόγου. Αυτά λοιπόν ε, σχετικά με την διάμεση επανεξέταση έχουν σχέση με τους στόχους έχουν σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αυτό μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να ε, ορίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι η προγραμματική περίοδος ε, αυτού του εργαλείου ξεκίνησε πριν από την έγκριση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε πώς όλα αυτά συμβαδίζουν με το διεθνές θεματολόγιο. Πρώτο λοιπόν σημείο της ενδιάμεσης επανεξέτασης ήταν να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο αντιπροσωπεία που να αφορά σε αυτό που αποκαλούμε εθνική στρατηγική στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε κατά πόσον οι διάλογοι και τα κονδύλια που προβλέπονται κατά πόσον όλα αυτά συμβαδίζουν με τα εθνικά προγράμματα. Ε, και επίσης και ε, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα. Γιατί ε, οι στόχοι αφορούν το να υπάρχει και μία κοινή πλατφόρμα. Σας λέω, όχι μόνο για να δαπανάμε χρήματα, αλλά επίσης και για να εξεταστούν τα βασικά στοιχεία τα οποία ε, καθορίζονται ως ε, ε, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βεβαίως, επειδή είναι κοινά τα προβλήματα, θα πρέπει να εξευρεθούν και κοινέ λύσεις. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Εμεί λοιπόν αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο τι περιγράφεται ως βασικό στοιχείο για να υπάρχει συνένεση, θεωρούμε βασικό στοιχείο είναι το φύλλο και η νεολαία. Βασικό είναι να, αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις, η βία κατά των γυναικών. Το ίδιο ισχύει και για τη νεολαία, δηλαδή πως κάθε χώρα προχωράει και τι ακριβώς θα κάνει έτσι ώστε να εξετάσει το θέμα της ανεργίας των νέων. Ε, έχουμε λοιπόν το θέμα των ε, βιώσιμων θέσιμων ανάπτυξης. Το τρίτο που είναι σημαντικό όσον αφορά τη συνένεση για τα πέντε πίτα αρχικά τα Peace, People, Planet και Prosperity στα αγγλικά, τα χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για να μπορούμε να αναλύσουμε σε ποιο βαθμό είμαστε με τις δικές τους τις προτεραιότητες και πώς ακριβώς αυτές οι προτεραιότητες ε, στηρίζονται από επρασανατολισμό του ε, προγράμματος ή ενδεχομένως από επιπρόσθετα κορδίλια. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι αυτή η ενδιάμεση επανεξέταση έχει περισσότερο με την ποσότητα και όχι με την ποιότητα. Γιατί σε επίπεδο αφομοίωσης ε, των κονδυλίων, εκεί εκτός από δύο-τρεις ε, περιπτώσεις δεν βρήκαμε ε, τραγικές περιπτώσεις όπου να πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν λειτουργεί και οπουδήποτε διαπιστώνουμε τέτοιου είδους καταστάσεις λειτουργούμε ανάλογα, δηλαδή συζητάμε με την άμεση ενδιαφερόμενη χώρα και ε, επαναπροσδιορίζουμε τη χρήση των κονδυλίων. Το ποσοτικό στοιχείο όλου αυτού ανέρχεται σε περίπου 5%. 5% αφορά την επανεξέταση. 5% λοιπόν καθορίζεται αφού πρώτα έχουμε εξετάσει ε, ποια είναι τα μεγάλα χάσματα σε σχέση με την απορρόφηση. Το 5% λοιπόν για να μπορούμε να επέμβουμε όπου κρίνεται απαραίτητο. Ε, Υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου εμφανίζονται βασικές ανάγκες και που δεν στηρίζονται από κονδύλια ε, που προβλέπονται για τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Ε, δουλεύουμε λοιπόν με αυτό το 5%. Θελήσαμε να το αναδιανύμουμε το 5% για να δούμε τώρα λιγάκι ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού, του διαλόγου και της, του αναπροσδιορισμού των κονδυλίων προέκυψε αύξηση του ποσού, ε, του τελικού ποσού που διατίθεται για τις επενδύσεις. Δηλαδή αυξήσαμε το σύνολο των κονδυλίων που διατίθενται για επενδύσεις. 667 εκατομμύρια ευρώ ε, από κοινού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το μέσο της αναπτυξιακής συνεργασίας και γι' αυτό το λόγο τα χρήματα αυτά ε, παραμένουν ε, στην περιφέρεια, αλλά ο τρόπος ε, με τον οποίο δαπανώνται χρησιμοποιώντα και τον πολλαπλασιαστή. Αυτό θα εξεταστεί. Πρώτα λοιπόν αυξάνονται τα κονδύλια ε, που προσφέρονται για επενδύσεις. Δεύτερον αυξάνονται τα κοντήλια για τις χώρες εκείνες ε, οι οποίες αντιμετωπίζουν την νόμιμη μετανάστευση και καθορίζουν ε, ε, και πολιτική ε, που προσανατολίζεται και στη μετανάστευση, που λαμβάνει υπόψη της στη μετανάστευση. Πολλές χώρες έχουν εξαντλήσει τα εθνικά κονδύλια και γι' αυτό λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι να τις βοηθήσουμε έτσι ώστε ε, να μπορούν μόνες τους να εκτελούν και τον προπολογισμό. Αυτά είναι ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Ένα τρίτο παράδειγμα ή αποτέλεσμα που θέλω να φέρω και έχει σχέση με τη μέθοδο που εφαρμόζεται και σε άλλους διαλόγους που γίνονται για τον φίλο άλλα παραδείγματα είναι να εντοπιστούν επιτυχημένες ε, παρεμβάσεις προς όφελος των γυναικών, ε, προς όφελος των εθνικών προγραμμάτων ε, προσπαθούμε σε κάποιες χώρες να προσφέρουμε επιπρόσθετα 5 εκατομμύρια που θα είναι ένα είδος επιβράβευσης για ειδικέ προσπάθειες που καταβάλουν ε, κυρίως ε, όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της διάστασης του φύλου. Αυτά είναι ε, η πολιτική που χαράσουμε σε σχέση με τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχει ένα περιθώριο του 5% που όμως ε, αυτό το 5% προσανατολίζεται κυρίως στις επενδύσεις και το υπόλοιπο στη μετανάστευση και στην κοινωνία των πολιτών. Αυτά όσον αφορά στο γεωγραφικό μέσο. Και κατόπιν αξιολογήσαμε ε, και τα ε, συγκεκριμένα θέματα του μέσου της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτά είναι συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν βέβαια γενικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Θέλω να σας πω ότι εκεί καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά λειτουργούν, ότι σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται στον στόχο για τον οποίο συστάθηκαν, ο στόχος παραμένει σε ισχύ. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι να προτείνουμε τη χρήση κονδυλίων με τέτοιο τρόπο που θα βοηθάει στο να συγκεντρώνονται πόροι για να στηριχτούν οι ευάλωτες χώρες για να στηριχτεί η ανθρωπιστική ανάπτυξη, να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών, ε, να διατεθούν περισσότερα χρήματα και κονδύλια για την ενίσχυση ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μεγάλων πόλεων θέλουμε να επεμβαίνουμε λιγάκι περισσότερο στο να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μεγάλων πόλεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον ε, αυτό είναι και ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο οφείλουμε να εξετάσουμε. Άρα δηλαδή πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις πόλεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη σημασία να αποδοθεί και στον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης, να σταθεροποιηθεί μια κοινωνία, να υπάρξει διαπολιτισμικός διάλογος. Μας ε, ενδιαφέρει να δίδονται κονδύλια και για την προστασία του ε, κλίματος και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με τη Συμφωνία COP21 στο Παρίσι. Επίσης, μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε και τον στόχο μας, ε, δηλαδή Όλα αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, τα θεματικά και τα γεωγραφικά. Δεν έχει προκύψει καμία σημαντική αλλαγή. Μας ενδιαφέρει να είμαστε καλύτερα εξεπλισμένοι για να στηρίξουμε καλύτερα τους ε, στόχους της ε, βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στην τελική φάση, είμαστε στην φάση όπου αρχίζουμε να ε, τα ε, πλαισιώνουμε όλα αυτά θεσμικά και πάνω σε αυτή τη βάση ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του 18 θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία γιατί αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω και βεβαίως με πολύ μεγάλη μου χαρά να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Απλώς για να είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα καλά. Αναφέρεστε σε ένα πρόγραμμα ενδιάμεσης αναθεώρησης για το γεωγραφικό πρόγραμμα του DCI και λέτε ότι θα δώσετε 5% του ε, χρηματοδότηση σε θέματα που αφορούν φύλλο, νεολαία, μετανάστευση, συμφωνία για την ανάπτυξη και επενδύσεις που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο για τις ε, θέσεις εργασίας στην Αφρική και για το θεματικό, ε, τις θεματικές ενότητες του Μέσου Αναπτυξιακής ε, Συνεργασίας δεν προτείνεται αλλαγέ. Για την πλευρά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης τι γίνεται, ε, ό,τι γίνεται και με το γεωγραφικό σκέλος του DCI, 5%. Ε, εφαρμόζεται δηλαδή ένα 5% και περιμένουμε λεπτομέρειες γι' αυτό μετά τα Χριστούγεννα και μετά θα υπάρχει χρόνος για να ελέγξουμε τι συμβαίνει. Ωραία. Συνάδελφοι, ο πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο Ερίκε Γκερερού. Παρακαλώ, Ερίκε. Ναι, ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα και δύο διαφορετικές διαδικασίες, αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση σχετίζεται με κάτι το οποίο έχουμε στη συνέχεια στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ανάπτυξης, μια έκθεση για την ε, εφαρμογή του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και ε, το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας. Προφανώ σε αυτή την περίπτωση αυτό το οποίο θα κάνει η Επιτροπή ανάπτυξη και αυτό θα το αναφέρω και αργότερα όταν θα συζητήσουμε το σημείο αυτό διότι θα είμαι και εισηγητή ε, για την έκθεση αυτή δεν πρόκειται τόσο για ενδιάμεση αξιολόγηση αλλά για μια αξιολόγηση για την εφαρμογή αυτών των μέσων και τρόπον την να δούμε πώς θα μπορούσαμε από πλευράς Επιτροπής Ανάπτυξης να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέσω πρόθεσμα για την αναθεώρηση των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών και την πιθανή αναδιάρθρωση ή μη αυτών των μέσων. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα ε, να ρωτήσω είναι ε, πόσες μπορούμε να έχουμε, πώς πληροφορίες μπορούμε να έχουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να έχουμε και στοιχεία για να κάνουμε τη δική μας την έκθεση, για να δούμε πώς λειτουργήσαν αυτά τα μέσα. Δεύτερον όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάποια πράγματα για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε θα υποβάλλετε την ε, γενική σας ανακοίνωση για τα πολιτές δημοσιογραμμικές προοπτικές 2020 και τη δημοσίευση κάθε μιας από των πολιτικών και των μέσων ε, για το μέλλον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι προς το παρόν η πρόβλεψη είναι η ανακοίνωση να γίνει το Μάιο. Δεν ξέρω αν όντω θα γίνει έτσι, αλλά αν είναι για το Μάιο... Ε, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα καλύψει όλο το 2018, όλο το 2019 και κατά πάσα πιθανότητα και ένα τμήμα του 2020 μέχρι να εγκριθούν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2020 και μετά και ε, να έχουμε και την τελευταία εκδοχή των τίτλων του προϋπολογισμού και των διαφόρων γραμμών. Αν όντως ισχύει αυτό θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε. Ευχαριστώ. Αρκετές ερωτήσεις. Ο κύριος ε, Ντέβα, ο αντιπροεδρός μας. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Μαρσελέση, για τις πολύ καλές παρατηρήσεις σας. για την επένδυσή μας για την Αφρική, την πρωτοβουλία για τις επενδύσεις για την Αφρική, στην οποία χρησιμοποιούμε και ε, χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να πάμε πέραν των 3-4 ε, δισεκατομμύριων μόχλευσης για να έχουμε τα 68 δις ε, στα οποία στοχεύουμε. Θα μπορούσαμε να πάμε πολύ πιο ψηλά για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο. Ε, ξέρω ότι ο κύριος Γιούνκερ επιθυμεί διακαώς να κάνει πολύ ε, ουσιαστική επένδυση στην Αφρική, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε σημαντικό αντίκτυπο με 30-40 δις, ε, μπορούμε με 200 δις. Αυτό σημαίνει να έχουμε πολύ περισσότερα κονδύλια μέσω μόχλευσης για να μπορέσουμε να έχουμε το δεκαπλάσιο ή το δεκαπενταπλάσιο της χρηματοδότησης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο. Ιδάλλως, ως συνήθως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εφευρικό ε, σχέδιο και να κάνουμε απλώς μια μικρή, ε, ένα μικρό θόρυβο. Ο κύριος Γκέρενς, Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαντσεβίζη κατά πόσον στον προβληματισμό του για το υπόλοιπο της περίοδου έχει συμπεριλάβει και το Brexit. Από ποια ημερομηνία και μετά θεωρείτε ότι δεν θα συνεισφέρει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο στον προπολογισμό και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας. Δεν είμαι βέβαιη κατά πόσο θα μπορέσει να απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριε Διευθυντά, σε ποιο βαθμό υποστηρίζω τα όσα κάνετε. Ε, υποστηρίζω, λοιπόν, και επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου, αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Καταρχάς, η πολιτική ε, ουσίας, που για μένα είναι το θεμελιώδες. Την παρατήρηση ε, του εισηγητή μας ότι δεν ήσασταν εκεί και λέ, λέτε, διαπίστωσα ότι εγώ ήμουν σκιώδης εισηγητής μια ώρα πριν έρθω στη συνεδρίαση, επομένως πρέπει να με ενημερώνετε. Και λέει εκεί ότι υπάρχουν κάποια ε, προβλήματα για τα καταπιστευματικά ταμεία και πρέπει να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο δωρητών και να υπάρξει συντονισμός. Το συζήτησα αυτό με τον Υπουργό Ασφαλείας και τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί είχαμε την ε, ημερομηνία, την ημέρα της ανεξαρτησίας και ε, αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμό σε επίπεδο κυβέρνηση. Το απάντησε και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλωστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Πολύ καλά και ωραία όλα αυτά. Αλλά συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, προφανώ. Ε, συμφωνούμε για το συντονισμό. Αν εσεί θέλετε να κάνετε συντονισμό σε επίπεδο κυβερνήσεων όλη τη βοήθεια και να σας δώσω και το σχετικό έγγραφο το οποίο δόθηκε, διότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα και πρέπει για τους στόχους που θέτουμε να γίνεται και ο συντονισμός των διαφόρων Υπουργείων, αλλά και των διαφόρων φορέων και των διαφόρων κονδυλίων. Και τα κονδύλια, όπως και το κονδύλιο για τις επενδύσεις, να προσαρμόζεται καταλήλως. Αλλά εσείς πρέπει να λάβετε τις αποφάσεις. Δεν μπορείτε να φοβάστε. Και δεν χρειάζεται να έρθετε καν. Το ακούσαμε πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και να σας παραπέμψω σε αυτό. Δεύτερον, να συμφωνήσω κι εγώ με τον συνάδελφο αναφέρεται και στα ιδιωτικά κονδύλια. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιαδήποτε βοήθεια η οποία δεν αφιερώνεται ε, στη δημιουργία πλούτου θα πρέπει να βοηθά στην ανεξαρτησία. Και αυτό σας το λένε όλοι όσοι ασχολούνται με την ανακτευσιακή βοήθεια. Η βοήθεια θα πρέπει να δίνεται για να υπάρχει πλούτος και ανάπτυξη επιτόπου. Αλλιώς είναι απολύτως αδύνατο να έχουμε οτιδήποτε. Και ευτυχώς που ε, συχνά οι Άγγλοι έχουν τόσο ρεαλιστική προσέγγιση, όπως επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ανάπτυξη στην Αφρική. Η βοήθεια ε, σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη βοήθεια. Ο δρόμος χρειάζεται συντήρηση για να μπορέσουμε να κάνουμε συντήρηση στο νοσοκομείο, για να πληρώσουμε την παιδεία, πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο. Αλλιώς θα χρειάζεται συνέχεια βοήθεια και θα γίνεται αένα αυτό το πράγμα. Δε... Ξέρω ότι είναι η φιλοσοφία σας αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τη δημόσια ενίσχυση και την ιδιωτική ενίσχυση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ Λίντα και να ευχαριστήσω και το Γενικό Διευθυντή για όλα όσα μας είπε, αλλά και για τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα επιτόπου. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι η πρώτη μου ερώτηση είναι αντίστοιχη με του συναδέλφου Ντέβα. Θα υπάρξει αύξηση των κονδυλίων πέραν αυτών των 3-4 δις, διότι αν αφαιρόμαστε σε 44 δις, τότε είναι λίγα τα ποσά. Ε, ακούσαμε πολύ συχνά και την είπατε εκπρόσωπο, την Φεντερίκα Μοντεγκερίνη, να λέει ότι κάθε χρόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, κάνουν ένα μαζικό σχέδιο. Βάζουμε όλα μαζί τα κονδύλια και φτάνουμε πάνω από 32 δις το χρόνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα 44 δις ε, για την ε, μόχλευση των 4 δις δεν αρκούν. Θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε κατά πόσον και τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να αυξήσουν τα κονδύλια. Διότι αν καταφέρουμε να υπερβούμε τα 200 δις, σίγουρα θα υπάρχει αντίκτυπος επιτόπου. Δεύτερη ερώτηση. Σήμερα γίνεται διάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η αναθεώρηση αυτή λαμβάνει υπόψη και το γεγονό ότι θα υπάρξουν πάρα πολλέ αλλαγέ τα επόμενα χρόνια. Ξεκινώντα από τη Συμφωνία του Κοτονού, θα υπάρξουν και άλλε αλλαγέ ε, ε, οι οποίε εφαρμόζονται στην Αφρικανική ε, επικράτεια, ε, η συμφωνία που θα υπογράψουμε του χρόνου με τα Ηνωμένα Έθνη και την πρόβλεψη για την ε, αποχώρηση των Ηνωμένων Εθνών ε, από την Παγκόσμια Συμφωνία για την Μετανάστευση, την οποία θα προσυπογράψουμε του χρόνου προφανώς ε, ε, δεν ε, έχει δεσμευτική ισχύ, αλλά πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία για τους μετανάστες, διότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς οδούς, αλλά επίσης να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και καταλήλως τη μετανάστευση. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κατάλληλο συντονισμός των κονδυλίων, χρειάζονται πόροι, και δεν ξέρω αν αυτό λαμβάνεται υπόψη και στην αναθεώρηση που γίνεται τώρα. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Να κάνω τότε εγώ ένα ερώτημα, να θέσω εγώ ένα ερώτημα σε σχέση με αυτό που είπε η Σισίλ έγκε 5% είπατε και έχουμε αυτήν την ε, μετάβαση στις προτεραιότητες. Πώς κρίνουμε την αποτελεσματικότητα κάποιων από των πολιτικών αυτών πριν μεταφέρουμε τα χρήματα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε για παράδειγμα τη Σύνοδο της Αφρικής και θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε να μας πείτε κάτι για την έκβασή της, γιατί εγώ δεν είδα κανένα σχετικό έγγραφο και οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί όλοι μου ζητούσαν ε, το σχετικό έγγραφο ενδεχομένω να μην είναι δική σα ευθύνη, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είναι εδώ η ΕΕΔ, το Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε, ήθελα να σας πω. Δεν ενημερώθηκε σωστά κατά διάρκεια της Αφρικανικής Συνόδου από την ΑΕΔ. Δεν λάβαμε καμία ενημέρωση ούτε την ε, Τετάρτη ούτε την Πέμπτη σε σχέση με τα αποτελέσματα της ε, Συνόδου. Είπατε ότι για αυτή την ενδιάμεση επανεξέταση ήρθατε σε επαφή με του εταίρου μα. Τι είπαν τι λένε για το να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη μετανάστευση. ο Γύρισα από τα Βιτζάν την ε, Πέμπτη, πάρα πολλές φορές ε, αναφέρθηκε η έκθεση για τα στρατόπεδα της Λιβύης είναι τεράστιο πρόβλημα για μας, για τους εταίρους μας και για την κοινή γνώμη εδώ. Πώς κρίνουμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα των ε, κονδυλίων για τη μετανάστευση πριν διαθέσουμε και άλλα ποσά σε τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Ευχαριστώ, Λίντα. Μπορώ να αρχίσω ενδεχομένω ε, με την ερώτηση του κυρίου Γκερέρο. Του κυρίου Γκερέρο. Το πρόβλημα που τίθεται γι' αυτό είναι ότι πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χώρος για να γίνει αυτό. Ο χώρος είναι να βρούμε τι μας λείπει προκειμένου να επιτύχουμε τα αποτελέσματα τα οποία από κοινού έχουμε αποφασίσει στην αρχή, δηλαδή την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, των SDGs είναι σαφές ότι θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση να ε, γίνει ένα ε, αμάλγαμα όλων αυτών. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα των προγραμμάτων, υπάρχουν συγκεκριμένα των πράγματα των μηχανισμών που υποστηρίζουν όλα τα προγράμματα, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη διαπραγμάτευση για τις πολιετήσεις δημοσιονομικού ε, προοπτικές που θα έχουμε στη συνέχεια. Προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο θα συνάδει και με το στόχο αυτής της διαδικασίας που καταρχάς είναι να εξετάσουμε κατά πόσο πόσον είναι ευστοχά και αποτελεσματικά τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Αυτό υπό τη στενή έννοια. Αν πάμε πέραν αυτών, ε, μπορεί να ξεκινήσουν συζητήσει που δεν έχουν πολιτικό πλαίσιο και επομένω επικεντρωνόμαστε σε αυτόν. Και για να προσθέσουμε και ένα περαιτέρω στοιχείο στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των μέσων, είπαμε ότι κανένας ε, μέσο δεν πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Βάση μιας αξιολόγησης επιπτώσεων, βάση και της γενικότερης αξιολόγησης, είναι αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης μέσων, ούτε το DCI, ούτε το Ταμείο Ανάπτυξης Βοήθειας, διότι κατά βάση συνάδουν και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και με όλα αυτά. Ε, και επιπλέον θα μπορούσε να ξεκινήσει και μια ολόκληρη συζήτηση η οποία ε, θα είναι σε ρήξη και με τη μελλοντική συζήτηση για τις πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία την οποία ε, κάνουμε με μια συζήτηση αρκετά περιορισμένη αν θέλετε, ταπεινή, γιατί έχουμε και μια διαδικασία που γίνεται με όλες τις χώρες του κόσμου και έχουμε και μια πολύ μεγάλη θεματολογία και αυτή η ανάλυση ε, ε, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρέπει ε, να έχουμε μέχρι 5%, διότι αν έχουμε κάτι πάνω από το 5% θα καταφέρουμε να έχουμε αντίκτυπο στις χώρες που δεν θα είναι απαραίτητος και θα είναι και αντιφατικό με την πραγματικότητα των όσων κάνουμε. Το πρόγραμμα παρουσίασης ε, των πολιετών δημοσιονομικών προεπτικών, όπω σωστά ανακοίνωσε ο κύριος Γιούγκερ, θα ε, γίνει ε, το Μάιο του 2018 και νομίζω ότι ο πρόεδρος είπε ότι καλό θα ήταν να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση όταν θα γίνει και το Brexit. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν αυτό, αλλά το σχέδιο είναι να παρουσιάσουμε τι προτάσει τις χρηματοοικονομικές προτάσεις για, το νέο, για τις νέες πολιτιετές δημοσιονομικές προοπτικές το Μάιο. Και ταυτόχρονα ή κάποιους μήνες αργότερα να έχουμε και την νομοθετική πρόταση. Ε, αυτά λοιπόν. Εγώ γι' αυτό θα αποφασίσω αυτό που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θεσμικό μου όργανο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Για τον ιδιωτικό τομέα, Νομίζω, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι ιδιαίτερα αφοσιωμένος σε αυτό γιατί δουλεύουμε πολύ σκληρά ώστε να υπάρχει το ε, επενδυτικό πλαίσιο ε, και εστιάζουμε στις διάφορες θεματικές ενότητες. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα από προγράμματα που λειτουργούν ε, για την κοινωνία των πολιτών, για την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απλώ για να πούμε ότι τώρα πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά και να αυξήσουμε ε, κάποιο άλλο, κάποια άλλη επένδυση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη και του ε, Μέσου Αναπτυξιακή Συνεργασία χρησιμοποιούμε αυτό το 5% για να γίνει μία αναδιάθεση. Αναφέρθηκα στα 600 κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε αυτό το τελευταίο τμήμα του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου για να αυξηθούν τα Όσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το, το, το, σχέδιο είναι να επιταχύνουμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη και επομένω αξιοπιστία για να ζητήσουμε περισσότερα στο επόμενο ΠΔΠ. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σα πω πόσα περισσότερα, αλλά δεν μπορώ να σα δώσω ένα αριθμητικό ποσό τώρα. Αλλά πάντως αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε αύξηση για να κάνουμε περισσότερα και να κάνουμε περισσότερα σε σχέση με το blending, αυτό το μείγμα. γιατί η εγγύηση, αν παραμείνει η ίδια, μπορεί να καλύψει περισσότερες επιχειρήσεις. Ε, είναι μικρά τα ποσά για την ώρα, αλλά νομίζω ότι είναι και σημαντικά παράλληλα. Ας μας δώσει, ας μας δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να αυξήσουμε την εμπειρία μας. Θέλω να τονίσω το εξή. Δεν μιλάμε γενικώ ε, για ε, εξωτερικές επενδύσεις. Μιλάμε για επενδύσεις που είναι υποφελείς για την ανάπτυξη και την, ε, την εξάλληψη της φτώχεια μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος μας ο βασικός. Κύριε Γκέρενς, ε, το Brexit ε, το έχουμε και δεν το έχουμε λάβει υπόψη. Δηλαδή, ναι, προφανώς είμαστε σε συνεργασία συνεχή και σε συζήτηση με τον Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος βλέπει τα πράγματα σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Δεν έχουμε λάβει υπόψη το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πληρώσει τα ποσά για τα οποία έχει δεσμευθεί. Δεν έχουμε έναν συντελεστή λοιπόν διορθωτικό στην υπόθεση κατά την οποία επί τη βάση διαπραγματεύσεων το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα θελήσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. ειδικά Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, είναι και μεγαλύτερε οι δεσμεύσει αυτέ, γιατί γίνονται σε διακυβερνητικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν ένα επιπλέον στοιχείο. Είναι σαφέ ότι παρακολουθώντα εκ του σύνεγγυ τι διαπραγματεύσει με τον κύριο Μπαρνιέ, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απτύξουμε σενάρια διαφορετικά. Αλλά όταν κάνουμε την ενδιάμεση επανεξέταση, νομίζω ότι πολιτικό και διαπραγματευτικό ε, δεν θα ήταν πολύ συνετό να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε το λογαριασμό που πρέπει να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία μείωση ποσών για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το Ταμείο Μπεκού και τα σχετικά καταπιστεύματα. Κοιτάξτε, εγώ τον Ιούλιο πήγα να είμαι υπεύθυνο ε, να είμαι ε, πρόεδρος της, του Στρατηγικού Συμβουλίου ε, ε, ο συντονισμός για το καταπίστευμα Μπεκού ε, ήταν πάρα πολλοί υπουργοί παρόντες των κέντρο αφρικανικών χωρών. Ό,τι κάνουμε λοιπόν, εντάξει δεν το καταφέρνουμε πάντα, προσπαθούμε να το κάνουμε και στα δύο ταμεία. Θελήσαμε να διαχειριστούμε ε, όσο το δυνατόν καλύτερα το Ταμείο Μπεκού ε, και για την Κολομβία. Έχουμε μια διαχείριση αποκεντρωμένη. Και γιατί θα το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να ενσωματωθεί στη συνεργασία με την ε, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Καλή είναι η συνεργασία, βέβαια χρήζει ε, ε, βελτιώσεως όπως πάντα, αλλά καλά πηγαίνει. Όσον αφορά τις επενδύσεις, περίπου το ίδιο πράγμα θα ήθελα να πω, επειδή μου μιλήσατε για δημόσια και ιδιωτική βοήθεια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για δημόσια βοήθεια, η οποία πρέπει να υποστηρίξει ε, όχι την ιδιωτική βοήθεια, αλλά τις ιδιωτικέ επενδύσεις. Γιατί, Γιατί λέμε ότι οι επενδύσεις που θέλουμε να διευκολύνουμε είναι αποδοτικές. Δεν κάνουμε επιδοτήσεις εμείς, ε, και κυρίως με την εγγύηση θέλουμε να έχουμε μια επιπλέον κάλυψη ε, ώστε ένας επιχειρηματίας που έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα αλλά έχει κάποια προβλήματα ίσως με την κυβέρνηση, τη διαχείριση που δεν είναι πάρα πολύ σταθερή ε, να μπορέσουμε κάπως να τον βοηθήσουμε. Αυτό όμως θέλουμε να κάνουμε, να διευκολύνουμε τις ε, εποφελείς ιδιωτικές επενδύσεις, τίποτα άλλο. Για το ερώτημα του σχεδίου Μάρσαλ ε, που μου κάνατε, που μου θέσατε. Κοιτάξτε, ε, τι εννοούμε. Ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή είναι 20 ε, δις περίπου διαθέτει στην Αφρική κάθε χρόνο. Είμαστε οι πρώτοι επενδυτές, άμεση επενδυτές, οι πρώτοι εμπορικοί εταίροι σε αγωγές-εξαγωγές και είμαστε και οι πρώτοι ε, ε, ας πούμε δημιουργοί εσόδων ε, Είμαστε λοιπόν μια πηγή εσόδων για την Αφρική πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, ώστε να μπορούν ε, οι ε, Αφρικανοί να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι ο τελικός στόχος. Τα κράτη-μέλη, το κατά πόσο ε, έχουν, είναι διαθέσιμοι. Κοιτάξτε, για το καταπίστευμα, για παράδειγμα, στη Βαλέτα είχαμε πει, ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε πει συγκεκριμένα, ότι τα κράτη-μέλη δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών οργάνων και αυτό το καταπίστευμα είναι κάπως μη εξισορροπημένο γιατί το ποσοστό συμμετοχή των κρατών μελών σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, είναι περίπου 10% η διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε και με την κυρία Γκρέσλε για αυτό το καταπίστευμα, αλλά προφανώ τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω και προσπαθούμε να πιέσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Η Ιταλία και η Γερμανία μετακινούνται κάπω, αυξάνουν τι εισφορέ του. Όσον αφορά τώρα την ε, αναθεώρηση των προγραμμάτων. Κοιτάξτε, αυτό είναι το σημείο εστίασης. Ε, θέλουμε, διατηρώντας μία αλφα σταθερότητα, γιατί δεν μπορούμε όλη την ώρα να ε, κάνουμε αλλαγές, με τους εταίρους αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε, ας αποφασίσουμε, ας συζητήσουμε ποιο είναι το σχέδιό σας σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Κάνουμε μια ανάλυση, βλέπουμε αν είναι χρήσιμο το πρόγραμμα, αν δεν είναι μπορούμε να το αλλάξουμε, αν υπάρχει υπερκατανάλωση μπορούμε να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. Αν υπάρχει υποαξιοποίηση, επειδή υπάρχουν κάποια κράτη που έδειξαν πάρα πολύ λίγο ενδιαφέρον, οπότε σε αυτή την περίπτωση σταματήσαμε την ε, ενίσχυσή μας και χρησιμοποιήσαμε αυτό το ποσό στο πλαίσιο του 5% για να καλύψουμε τις χώρες οι οποίες ε, μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα ποτά. Τώρα, πώς ε, κρίνουμε την αποτελεσματικότητα. Ε, βάσει των αποτελεσμάτων επιτόπου χρησιμοποιούμε τους ίδιου δείκτες. Δεύτερον, όταν υπάρχει υποστήριξη του προπολογισμού, ε, ε, υποστήριξη προπολογισμού ε, είναι, πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αποτελέσματα. Όταν υπάρχει η μακροοικονομική προσπάθεια να υπάρχει ένα μακροθόμενο αποτέλεσμα ή ένα, μία δόση μεταβαλλόμενη ανάλογα με το αποτέλεσμα επιτόπου, νοσοκομεία, οδικοί άξονες κλπ. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ένα είδος βαθμονομημένου πίνακα που το οποίο χρησιμοποιούμε επίση στο ποσοτικό κομμάτι, πόσα χρήματα διατίθενται. Όσον αφορά τη μετανάστευση τώρα, εντάξει είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρό και δικαίω υπάρχει το βραχυπρόθεσμο, ε, το οποίο είναι ουσιαστικά ανάπτυξη υποδομών των κρατών μελών ε, και την αντιμετώπιση ε, του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Να πάρουμε για παράδειγμα την, ε, οδό της κεντρικής ε, Μεσογείου, εντάξει τόσοι άλλος θα μιλήσετε και για τη Λιβύη πιο μετά. Η συγκεκριμένη οδός έχει δει μια πολύ σημαντική μείωση κίνησης και φυσικά έχει πληγεί και η οικονομία όλων αυτών που ασχολούνται με αυτήν την οδό σε μερικές περιπτώσεις όμως υπάρχει πολύ πιο ε, παρεμβατική ας πούμε συμμετοχή την οποία μπορούμε και φυσικά να ε, ποσοτικοποιήσουμε σε αποτέλεσμα πολύ πιο συγκεκριμένα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση όπως το Μάλι για παράδειγμα αν λαμβάνει ένα top-up, ένα επιπλέον ποσό γιατί έχει χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό, έχει δείξει προθυμία αλλά και ικανότητα αξιοποίησης περισσότερων, περισσότερων και από κοινού αποφασίζουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε το Μάλι όχι μόνο στα σύνορα, γιατί με το Μάλι νομίζω ότι είμαστε παρόντες, αλλά και διαχείριση άλλων πτυχών, όπως για παράδειγμα την απουσία του κράτους στην εκπαίδευση συγκεκριμένα, που είναι ένας από τους βασικούς τομείς, στους οποίους ε, η τρομοκρατία στο κεντρικό Μάλι και η φτώχεια συνδυάζονται, ώστε να οφείται ο κόσμος στην τρομοκρατία. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να τους πούμε, συμφωνείτε με αυτή την ιδέα, αν συμφωνείτε υπογράψτε. Εντοπίζουμε λοιπόν μια καλή μέθοδο και καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Μερικές φορές δεν συμφωνούμε με κάποιες χώρες ε, για τις οποίες αποφασίσαμε ή προτείναμε τέλος πάντων να κόψουμε τη βοήθεια, δεν ε, είναι ικανοποιημένες άλλες, δεν είδαν τα ποσά τους να αυξάνονται δεν είναι κάτι ε, το οποίο ικανοποιεί όλο τον κόσμο, αλλά είμαι ότι γίνεται με έναν δίκαιο τρόπο ε, και συνεργαζόμαστε μαζί τους, μιλάμε μαζί τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε λοιπόν τι περικόπτεται και, τι, και πού πηγαίνει. Χάιντι Χάουταλα. Μπορείς να κάνεις την ερώτηση τώρα, ναι. Δυστυχώς ε, έπρεπε να λείψω για ένα τέταρτο και ξέρω ότι είχατε μια ανταλλαγή απόψεων, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω λιγάκι σχετικά με το τι πιστεύετε για αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ε, αφρικανικές ε, κυβερνήσεις και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Διότι βεβαίως πρέπει να πω, εκπλαγήκαμε πάρα πολύ που αρκετές ημέρες πριν από συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ε, που έλαβε χώρα στο Αμπιτζάμπι. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα μετάφρασης, αλλά δεν έχουν ακόμα δοθεί τα κείμενα, κανένα κείμενο. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι ότι οι αφρικανικές κυβερνήσεις δεν τάσσονται τόσο πολύ υπέρ του ρόλου που μπορεί να παίξει η κοινωνία των πολιτών. Αυτό όμως είναι πρόκληση για μας, γιατί στη δική μας την άποψη περί πολιτικής είναι απαραίτητο να υπάρχει διάλογος με την κοινωνία των πολιτών σε όλους τους τόνους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει. Άρα δηλαδή θέλω να ρωτήσω υπάρχει κάποια δυνατότητα να τους πείσετε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στην κοινοβουλευτική συνέλευση που είχαμε η πρόεδρος μας, η κυρία Κίνγκε και πολλοί άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να ρίχνουμε μονίμως το βάρος στους άλλους, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και η δική μας ευθύνη είναι να δώσουμε το καλό παράδειγμα με την σωστή διακυβέρνηση και αυτό είναι και το μήνυμα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από εσάς ε, τι πιστεύετε εσείς ε, σχετικά με αυτή την προτιμία, έστω τουλάχιστον κάποιον, τουλάχιστον κάποιον στην Αφρική. Και μήπως μπορείτε και να μας ενημερώσετε και για την ε, συζήτηση που είχατε με τους νέους από το, την ακτή Ελεφαντοστού, από νέους δηλαδή οι οποίοι επέστρεψαν από τη στη Λιβύη μάλλον από τη Λιβύη στην ακτή του Ελεφαντιστούν. Ε, δεν έχουν εκεί προοπτικές ε, και αυτό βέβαια είναι μόνο μία χώρα στην περιοχή. Ε, ακόμα και αν είναι κανείς επαγγελματίας, δεν έχει δουλειά. Ε, δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι το καθήκον μας ε, να στηρίξουμε τις αφρικανικές χώρες και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αυτό είναι μια Ηράκλεια πρόκληση. Βεβαίως δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε για αυτούς, αλλά μπορούμε να τους στηρίξουμε στο να το επιτύχουν αυτοί αυτό. Πολλοί ζήτησαν να υπάρξει πραγματικός ε, διάλογος και όχι ο ένας να ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον. Νομίζω ότι ως βουλευτές ε, οφείλουμε αυτά τα θέματα, αυτό το θέμα να το προάγουμε. Ε, όσον αφορά το Αμπιτζάμ, ε, είδαμε ότι εκεί στο Αμπιτζάν ε, έξω από την πρωτεύουσα έχουμε ακόμα σλάμ ε, δεν υπάρχει ικανοποιητική ανάπτυξη. Ξέρω ότι πρέπει να πάτε και σε άλλη επιτροπή. παρακαλώ σύντομα. Ναι, συγγνώμη κύριε Διευθυντά, η απάντησή σας δεν με ικανοποιεί και γιατί αυτό. Διότι δεν είναι το ίδιο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το συντονισμό και καλεί ε, τον Υπουργό από την κυβέρνηση η οποία με ένα ad hoc τρόπο, χωρίς θεσμική ε, διαδικασία, συστήνει μία επιτροπή συντονισμού όπου ε, καθορίζει κάποια πράγματα για τους δικούς τους στόχους επιβίωσης, διότι περί επιβίωσης πρόκειται. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, διότι δεν είναι ένα και το αυτό αυτά τα πράγματα. Ναι, ευχαριστώ. Αν ε, μπορώ να απαντήσω, ζητώ συγγνώμη, μπορεί να μην εκφράστηκα σωστά. Εγώ δίνω παράδειγμα. Ε, οι υπουργοί που βρίσκονται στην Επιτροπή είναι ακριβώς ε, ένα παράδειγμα ότι υπάρχει ένα επιπλέον εργαλείο για να γίνει συντονισμός. Αλλά γνωρίζετε ότι οι κεντροαφρικανικές κυβερνήσεις με τη δική μας τη χρηματοοικονομική υποστήριξη έχουν συστήσει μια επιτροπή η οποία θα ε, εξετάσει τα προγράμματα τα οποία θα υποβληθούν από εκεί και πέρα στους εταίρους ε, και σε αυτούς οι οποίοι δίνουν τα κονδύλια. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να συντονίσουν τη βοήθεια. Εμείς βοηθούμε αλλά αυτοί πρέπει να αναλάβουν τη, τη, τη σκητάλη. Συγγνώμη αν δημιούργησα κάποιες αμφισημίε, αλλά αυτό ακριβώς εννοούσα. Όσον αφορά τη σύνοδο, στην τελική ανακοίνωση που είδα στο τέλος, το αφήνω και στο συνάδελφο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αν έλεγε και κάτι άλλο, ε, πέραν της μετάφρασης που διάβασα εγώ, μπορώ να σας πω το εξής. Η σύνοδος αυτή, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, ε, διότι συμμετείχα και σε όλες τις συνόδους και έχω και μια αίσθηση του πώς ε, πάνε τα πράγματα, είναι μια σύνοδος με ένα καλό αποτέλεσμα αλλά και μιας κάποιες μορφής μετάβαση. Η αλλαγή νοοτροπίας, η αλλαγή σχέσης ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μια νυχτή. Ε, υπήρξε μια στιγμή καλή συζήτηση και αυτό δείχνει ότι λαμβάνουμε ένα τον άλλο σοβαρά υπόψη και αυτό δεν μεταφράζεται στο κατά πόσον είχαμε αμέσως αυτά αποτελέσματα ε, δεν είχαμε από όλε τι πλευρέ, για παράδειγμα, ο περιβόητο αυτό κατάλογο των προγραμμάτων τα οποία επρόκειτο να εγκριθούν στη Σύνοδο ω ε, ε, προσάρτηση στα συμπεράσματα δεν εγκρίθηκε τελικά. Γιατί? Γιατί μετά από τη συζήτηση και οι δύο πλευρέ θεώρησαν ότι πρέπει να γίνει κάτι επιπλέον πέραν ε, των όσων ήθελαν να κάνει κάποιο στο αφρικανικό σκέλος. Ήθελαν δηλαδή μια λίστα με τα ποσά του τι θα δίνουμε και κάποια πράγματα που δεν θέλαμε εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε. Δεν θέλαμε να έχουμε να θα πάρετε τόσα, αλλά θέλαμε έναν προσανατολισμό. Ε, και αυτό φυσικά σημαίνει ότι δεν έχουν τελειώσει αυτά, εκκρεμούν. Μία ακόμα εκκρεμότητα, επί της οποίας όμως έχουμε συμφωνήσει, είναι ότι τώρα το συντομότερο δυνατό πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα μνημόνιο συνεννόηση ε, για τις σχέσεις ειρήνης και σταθερότητας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα το έχουμε στα παραδοτέα έγγραφα, αλλά η σύνοδος και η συζήτηση που προέκυψε κατέδειξε ότι πρέπει να το επεξεργαστούμε λίγο περαιτέρω. Και στις δύο όμως περιπτώσεις, τα θέματα επί των οποίων συζητούσαμε αναγνωρίστηκαν πλήρως. Δηλαδή, ε, υπάρχει μια μηδέα αναγνώριση των αλλαγών που δημιουργούν ίσως και κάτι επιπλέον στην ατμόσφαιρα και δίνουν μια αίσθηση ότι δεν υπήρχε πλήρη συνένεση. Αλλά μεταξύ μιας ατμόσφαιρας πλήρης συνένεσης που βασίζεται απλώς σε κάποια ε, ε, γραπτά πράγματα τα οποία διαβάζουν και μια καλή ανταλλαγή απόψεων υπάρχει διαφορά και ήταν τελικά τα αποτελέσματα. Και όσον αφορά την τελική δήλωση θα σας τα πει στον συνάδελφος, αλλά υπήρχε δήλωση. Αυτό που είπα και είναι και κοινό μυστικό, είναι ότι από αφρικανική σκοπιά υπήρχε κάποια δυσκολία στο συντονισμό. Εμεί από πλευρά μα, ε, ξέρετε, με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η Γενική Διευθύνση ΔΕΦΚΟ ήταν προετοιμασμένοι και υπήρχε συντονισμό. Υπήρχε προφανώ μια πολύ πιο σύνθετη κατάσταση από πλευρά του. Ε, τα έγγραφα λοιπόν καθυστέρησαν, η δυναμική μεταξύ τους ε, πρέσβης ε, και μεταξύ των πρέσβεων και των επιτροπών φάνηκε ότι δεν είναι τόσο εύκολη. Υπήρχε κάποια δυσκολία συντονισμού που κατέδειξε ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα θέματα της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαία, από τη μια φάνηκε να υπάρχει ε, ένα επίμεχο ζήτημα, αλλά τελικά δεν ήταν. Ε, ε, υπάρχει ανάγκη δηλαδή να θέσουμε σε λειτουργία ένα περιβάλλον το οποίο θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Το θέμα της κοινωνίας είναι πάντα σε όλες αυτές τις συνόδους σημαντικό, διότι πάντα υπάρχουν οι δύο πλευρές επιχειρημάτων, η μια λένε ότι, ότι διαλέγετε αυτό που σας αρέσει και δεν διαλέγετε αυτά που δεν σας αρέσουν. Πάντα έτσι γίνεται. Στη δήλωση όμω υπάρχει αναγνώριση των όσων κάνουμε με την κοινωνία των πολιτών, με την νεολαία, με τις τοπικέ αρχές, αν θυμάμαι καλά τη διατύπωση και το καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι έτσι πάνε τα πράγματα. Τώρα για τους ε, ε ανθρώπους από την ακτή του Ελεφαντοστούν που επαναπατρίστηκαν από τη Λιβύη, ε, ξέρετε ότι υπήρχε μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, και άλλων εταίρων για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στη Λιβύη. Προσπαθούμε να δράσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα και κοιτάμε να δούμε πώς ε, και πού μπορούμε να έχουμε ένταξη και υπάρχει κάτι το οποίο πάντα υπερασπίστηκα εδώ και κάποιες φορές επικρίθηκα και γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η σχέση με την κοινωνία των πολιτών και του Οργανισμού Μετανάστευσης που λαμβάνει υπόψη του αυτούς που επιστρέφουν. Είτε επιστρέφουν θελοντικά, είτε επιστρέφουν υποχρεωτικά, που επιστρέφουν από τη Λιβύη, από την Ευρώπη. Κάπου φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να τους φροντίσουμε. Αν δεν τους φροντίσουμε θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Τώρα, στην ακτή του ελεφαντιστού ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να νιώσουν ότι δεν έχουν ευκαιρίε. Αυτό το γνωρίζουμε όμω. Γι' αυτό προσπαθούμε να του βοηθήσουμε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να έρθουν στη θέση εργασία, να συστήσουν μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αλλά θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται. Προσπαθούμε να τους φροντίσουμε ε, άμα τη επιστροφή τους, διότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες, αλλά ε, υπάρχει και ε, εχθρικότητα από τις κοινότητές τους, διότι έχουν επενδύσει σε αυτούς για να προσφέρουν κάτι καλύτερο και πολλές φορές απογοητεύονται από αυτούς. Ε, και αυτό είναι και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα το έχουμε και μαζί μας για πολύ καιρό. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα όμως φαίνεται ότι κάποιοι έχουν αφυπνιστεί στη Λιβύη, δεν είναι καινούργια διαδικασία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το επόμενο θέμα ε, που θα εξετάσουμε είναι για τη Λιβύη και θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε. Η κυρία Ντεμπέργκ, δεν ξέρω, είναι παρούσα. Δεν ξέρω αν θέλετε ή μπορείτε να μας μιλήσετε για την δήλωση ε, τη συνάντηση κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Υπάρχει κάποιο που να μπορεί να τοποθετηθεί από αυτού. Ε, εντάξει, μπορείτε να μιλήσετε εσεί ε, και μετά να μιλήσει η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, διάμεση αναθεώρηση του αναπτυξιακού μέσου, όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής, αυτή η όλη η πράξη γίνεται σε συνδυασμό δεν ρωτάω αυτό. Εγώ ρώτησα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί τη συζήτηση την είχαμε ήδη. Και έχουμε ένα άλλο σημαντικό θέμα και έχουμε καθυστερήσει. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καλώς. Δεν χρειάζεται τώρα όμως να πείτε και πάλι τα ίδια. Ένα πράγμα θέλω να υπογραμμίσω, τη σημασία του διαλόγου ο οποίος έλαβε χώρα ανάμεσα στις αντιπροσωπείες και με κάθε τοπικό ε, εταίρο σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, στα αποτελέσματα φαίνεται ο διάλογος που έλαβε χώρα. Αυτό ήθελα να πω. Και όσον αφορά την ερώτησή σας για το έγγραφο από αυτή την συνάντηση κορυφής, Δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σα. Ε, παρακαλώ μήπως υπάρχει κάποιο από την Υπηρεσία εξωτερική δράση που να μπορεί να απαντήσει. Αν όχι τότε να το διαβιβάσετε ότι ε, δεν έχουμε αυτό το έγγραφο. Το παλεύουμε, το προσπαθούμε εδώ και καιρό αλλά δεν το έχουμε και θέλουμε να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι και θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε άλλα δύο σημαντικά θέματα που ακολουθούν και έχουν βέβαια με το ίδιο θέμα. Είναι το σημείο υπαριθμών 8. Πρόκειται για την εφαρμογή του Μέσων Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτά θα μας βοηθήσουν στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση, στις προετοιμασίες για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε δύο μιλητές από την Concord και από την Voice. Έχουμε και τον εισηγητή κοντά μας, τον κύριο Γκερέρο. Θέλετε εσείς να μιλήσετε πρώτος ή να μιλήσουν οι άλλοι, Ενρίκε. Να μιλήσουν πρώτα οι δύο προσκεκλημένοι και μετά ε, θα λάβετε εσείς το λόγο, γιατί... Ε, πραγματικά δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα ακολουθήσει η διάλογος. Άρα δηλαδή θέλουμε να δούμε πόσο καλά έχουν προχωρήσει τα προγράμματα και χαίρομαι πολύ που έχουμε κοντά μας την κυρία Βερνό εκ μέρους της ε, Concord που θα μας μιλήσει υποθέτω Μάλλον και οι δύο θα μιλήσουν για το μέσο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Από την Κονκόρτ έχουμε την κυρία Ίνκη Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει πρώτος. Η κυρία Βερνό θα μιλήσει πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας προσωπήσω εκ μέρους της ε, Concord. Είναι πολύ σημαντική ευκαιρία για να δούμε ε, κατά πόσον τα ε, μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας εξακολουθούν να εξυπηρετούν το στόχο. Και θέλω επίσης να σας ε, ενημερώσω και για τον προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης και για τα βασικά στοιχεία για το επόμενο σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Να σας πω κάποια στοιχεία ε, που αφορούν στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, θα εστιάσω σε ορισμένα βασικά θέματα και ελπίζω αυτά να είναι και χρήσιμα γιατί θα τα εντάξετε και στον διαρθρωμένο διάλογο. Ε, θα μιλήσουμε για το DCI, για το μέσο της αναπτυξιακής συνεργασίας και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ακόμα βέβαια είναι πολύ νωρίς ε, για να εξάγουμε συμπεράσματα. Και θα μιλήσω και για τα βασικά στοιχεία. Ε, σύντομα ελπίζουμε να ε, ανταλλάξουμε απόψεις για περισσότερα θέματα, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τα βασικά στοιχεία. Είμαστε μια πλατφόρμα 28 κρατών. Όλα αυτά απαιτούν μεγάλο συντονισμό και ε, με μεγάλη χαρά να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, να δούμε λιγάκι την υποστήριξη που παρέχουμε ε, Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, αλλά αυτό που επίσης ε, απαιτείται είναι να γνωρίσουμε και την προστιθέμενη αξία των των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ε, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλες οργανώσεις ε, κοινωνίας ε, των πολιτών. Οι κοινωνίες των πολιτών διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλληλοσυμπλήρωση. Όσον αφορά το Παναφρικανικό πρόγραμμα, αυτό είναι αρκετά περιορισμένο και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ε, εκεί ε, έχουμε μόνο το 60% των ΝΙΠ και επίσης ε, θα ήταν καλό να έχουμε και περισσότερα ε, εθνικά προγράμματα. Ε, επίσης υπάρχουν και διάφορα επίπεδα υποστήριξης. Έχουμε τρεις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες ε, δεν έχουν συγκεκριμένους φακέλους. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει παντού υποστήριξη ε, στο, ε, στις οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών. Γιατί όπως αναφέρεται και προηγουμένως, δεν υπάρχει πλέον αρκετό περιθώριο για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό λοιπόν πρέπει να προκύψει ως προστιθέμενη αξία. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και αυτά εξαρτώνται και από την ε, Concord, η οποία έχει ε, υποβάλει μία συγκεκριμένη έκθεση, ε, προσπαθεί να δείξει πώς ακριβώς λειτουργούν οι οργανώσεις κοινωνίας των πελητών επιτόπου. Άκουσα ότι υπάρχει κάποιο συντονισμός για τις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά εξακολουθεί και εκεί να υπάρχει ανάγκη συντονισμού και προγραμματισμού οι, κοινωνίες, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ε, πρέπει να ενταχθούν στο Παναφαρικανικό πρόγραμμα. Ε, ακόμα δεν υπάρχει πλήρη, ε, πλήρης συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολο του προγράμματος. Όσον αφορά τα νέα βασικά στοιχεία, εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ισότητα των δύο φύλων τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα στην μετάφραση αφορούν ε, ε, στο ότι ε, δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Άρα δηλαδή εκεί τα πράγματα μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα. Και αν δούμε το EDF, κάναμε μία ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων. Σε όλα αναφέρεται το θέμα του φύλου, αλλά μόνο σε ένα πρόγραμμα υπάρχουν τα κονδύλια για να στηριχθεί η ισότητα των δύο φύλων. 19 είπαν ότι το κάνουν αυτό ε, σε βασικούς τομείς, αλλά δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα. Ακούσαμε προηγουμένως ότι θα υπάρξει αύξηση των κονδυλίων 50 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, και Επίσης ε, αναφέρθηκε και μία πρωτοβουλία που ε, ανελήφθη ε, το Σεπτέμβρη. Εμείς τη χαιρετίζουμε, αλλά θέλουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τα επιπρόσθετα κονδύλια για την ισότητα των δύο φύλων. Όσον αφορά την χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, εκεί πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και επίσης να βελτιωθεί και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών ο συνάδελφός μου ήταν ε, στην συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Σε εμά δεν δόθηκε η δυνατότητα να παρέμβουμε στη συνάντηση κορυφής. Καλό είναι που θα υπάρχει αυτή η διακήρυξη, αλλά εμείς δεν μπορέσαμε να παρέμβουμε. Ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά για να γίνουν και βλέπετε ε, στο πρόγραμμα ότι γίνεται συνεχώς λόγος για τη δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δει κανείς ε, το EDF, EDF ε, και τα εθνικά προγράμματα, τα NIP, θα μπορούσε να προβληθεί περισσότερο η χρηστή διακυβέρνηση. Ένα άλλο θέμα είναι η νεολαία Ε, που αυτό ε, παίζει σημαντικό ρόλο και είναι καλό, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά αποτελεσματικά. Θέλω να σε επισημάνω το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σχεδιασμός ε, στο σχεδιασ... να υπάρχει σχεδιασμός στις θέσεις απασχόλησης που αφορούν στους ε, νέους. Αυτό το θέμα το θίξαμε και στην Επιτροπή. Και όσον αφορά ε, την ανθρώπινη συμπερίληψη, ε, αυτή τη διάσταση, με βάση την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2015 ήμασταν στο 21%. Ε, αν δει όμως κανείς τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, εκεί δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία, κανένα σημαντικό ποσοστό. Αν δει κανείς τα εθνικά προγράμματα, ε, βλέπουμε ότι μόνο το 14% έχει σχέση με την ε, κοινωνική και ανθρώπινη συμπερίληψη. Τα, όλα, τα υπόλοιπα αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά στη διάρκεια των ετών, όχι μόνο για μία χρονιά, για το 2015. Το ίδιο ισχύει και για την κλιματική αλλαγή. Ε, σας είπα ότι ένας από τους στόχους ε, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έχουμε τις ε, προκλήσεις, τις ε, δημόσιες προκλήσεις. Στην ε, πρακτική βλέπουμε όμως ότι υπάρχει κατακαιρματισμένη προσέγγιση. Άρα μπορούν να γίνουν περισσότερα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και τέλος, όταν μιλάμε για ανάμιξη, για τα καταπιστευματικά ταμεία, για τα μείγματα και για τα καταπιστευματικά ταμεία, δεν είναι και τόσο ναι, αυτά, αλλά εμείς θέλουμε να επενθυμίσουμε ότι δεν θα πρέπει αυτά να είναι εις βάρος των αρχικών στόχων. Για μας είναι απόλυτα σαφές ότι θα πρέπει κανείς να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι στόχοι και πρώτα να ξεκαθαρίσει και ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Η ισορρευτικότητα είναι σημαντική, εφόσον ή όταν υπάρχουν ήδη μηχανισμοί blending, ε, πρέπει να δούμε ε, κατά πόσον ε, οφείλουμε να επιμείνουμε σε αυτό. Και εδώ πάλι είναι σημαντικό να υπάρχει μία αξιολόγηση εκ των προτέρων. Και ό,τι χρησιμοποιείται για αυτό το μηχανισμό ανάμιξης θα πρέπει να ακολουθεί και τις προδιαγραφές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τώρα όσον αφορά την ατζέντα ε, της Μπέμπα, ε, εκεί προφανώς πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, αλλά το θέμα δεν είναι κατά πόσον θα υπάρχει ο στόχος ε, της συνεργασίας. νομίζω ότι ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει στρατηγική συμμετοχή να έχουμε κατά νου τις ανάγκες των ανθρώπων όταν σχεδιάζουμε αυτά τα προγράμματα. Για τα καταπιστευματικά ταμεία έχουμε πέντε, εντυπωσιακό αυτό, και βεβαίως κατανοούμε γιατί κάποια συστάθηκαν, αλλά παράλληλα θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας να πούμε ότι ένας στόχος είναι ότι αυτά δεν πρέπει να συνδέονται με τα εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Επίσης, ε, να έχουμε κατά νου ότι αυτά τα ε, καταπιστευματικά ταμεία ε, θα πρέπει να προσφέρουν προσθέμενη αξία, όχι απλά επικάλυψη. Και κάτι το οποίο συζητήθηκε επίσης είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ε, σε κάποια ταμεία, ούτε και πώς συστήθηκαν, ούτε και πώς ακριβώς λειτουργούν. Είναι εργαλεία ε, που είναι πολύ ευέλικτα, αλλά η διαδικασία δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που έχουμε. Ε, αυτά με λίγα λόγια για την διάμεση αναθεώρηση και όπως βλέπετε ε, μπορούμε αρκετά να μάθουμε ε, βασικές αρχές που πρέπει να ισχύουν ε, σχετικά με το επόμενο σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, τα βασικά στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε σε ένα έγγραφο που θα σας δώσουμε πολύ σύντομα. Αλλά το βασικότερο μήνυμα που θέλουμε να σας μεταφέρουμε σήμερα είναι ότι όταν θα περάσουμε στα επόμενα αναπτυξιακά μέσα ανεξάρτητα από τον προπολογισμό, για μας αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμους στόχους. Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι καθοριστική σημασία για μας. Δεν θέλουμε <laughs> να ε, υπάρχει κίνδυνος, αλλά να υπάρχει σαφής ε, διαχωρισμός. μέσα τα οποία δεν μπορούν να επιλεγούν, να υπάρχει αυτή διαχωρισμός από τα επιλέξιμα. Θέλουμε να υπάρχει κοινοβουλευτική εξέταση και όσον αφορά τη χρηματοδότηση θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αύξηση της επίσημη αναπτυξιακή βοήθειας, τουλάχιστον να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο και προφανώς θα ζητήσουμε αυξημένο προπολογισμό. Όσον αφορά τώρα τους συλλογικούς, ε, ε, το συλλογικό στόχο του 0,2% ε, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, θεωρούμε ότι εκεί μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εστίαση συγκεκριμένα ως προς τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο αυτό του 0,2% Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για την κάλυψη των βασικών στόχων, να μην μειωθεί ο προπολογισμό, συνδιαχείριση ε, και μακροχρόνιο προγραμματισμός. Και όταν φτάνουμε τώρα στο στην τελευταία αρχή, θα θέλαμε η βαθμονόμηση που υπάρχει για την ανάπτυξη και την, ε, τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, αν είναι δυνατόν να έχουμε μία αύξηση ε, του, της τάξης του 50% και 20% του ε, ΑΕΠ αύξηση ε, για τις στοχευμένες δράσεις. Όπως είπαμε, ε, πρέπει να υπάρξει μία προχρηματοδότηση και κοινός προγραμματισμός ε, με κάποια συμμετοχή των κρατών μελών. Και κάτι ακόμη είναι το θέμα της ευελιξίας ε, έναντι της προβλεψιμότητας ε, συγγνώμη, διακόπτη Πρόεδρο, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα μελλοντικά προγράμματα για κάποια άλλη στιγμή. Για την εφαρμογή των ε, υφισταμένων προγραμμάτων θέλουμε να μιλήσουμε. Α μην ε, αγωνιούμε τώρα για τα μελλοντικά. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μα μέχρι να αρχίσει αυτή η συζήτηση. Μην ανησυχείτε, θα το ξανασυζητήσουμε. Μπορεί να διαβάσουν ε, μόνοι του τι διαφάνειε οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να σα διακόψω δυστυχώ η κυρία Μπρίς τώρα από τη Voice ε, που εκπροσωπεί τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Ε, για να δούμε λοιπόν την χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, για τα ανθρωπιστικά προγράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς τι κάνουμε. Ε, θέλαμε να μεταγράψουμε τους στόχους ε, της συνθήκης Λισαβόνας ε, που έλεγε ότι οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετεραιότητας και της μη διάκρισης. Μα ζητήθηκε λοιπόν να προβληματιστούμε επί των τριών αυτών στοιχείων, της απόδοσης των ανθρωπιστικών μέσων, της βελτιώσης και την ανθρωπιστική νομοθεσία. Να αρχίσω με το πρώτο. Ε, πόσο, πόσο καλά έχει το ανθρωπιστικό μέσο λειτουργήσει. Η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος πολλές φορές δίνει τη δυνατότητα να δούμε τι μεγάλες καινοτομίες χρειαζόμαστε, τι δεν λειτουργεί καλά και να δούμε με τι λειτουργεί καλά. Και από αυτό θα ε, ξεκινήσουμε. Αυτό που μας αρέσει στην ΕΚΟ και στο ανθρωπιστικό μέσο. Είναι, γνωστή, ο, είναι γνωστό ότι δεσμεύεται από και, και, και σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό ανθρωπιστικό δίκαιο ε, και αυτό, σημαίνει, αυτό, αυτό σε αντίθεση με πολλά άλλα ε, κράτη-μέλη που έχουν πολύ πιο πολιτικοποιημένες και μεροληπτικές αποφάσεις. Βασίζεται λοιπόν ε, σε ξεχασμένες κρίσεις τις οποίες προσπαθεί να φροντίσει και βάσει αναγκών επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό το ανθρωπιστικό μέσο πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, καθοδηγείται από ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο πολιτικής. Νομίζω σε αυτήν την ε, ε, αίθουσα μιλήσαμε για την πλήρη συνένεση ε, ως προς το, την, διατήρηση αυτή του ανθρωπιστικού μέσου, γιατί είναι ένα κοινό παρονομαστής ε, είναι ένα ρεαλιστικό έγγραφο ε, και τα αποτελέσματά μας πρέπει να βασίζονται σε αυτό, όπως είπε και ο κύριος Γκερέρο Σαλόν. Δεν είναι ένα, ε, ένα απλό μέσο, είναι ένα μέσο που πρέπει να συνδυάζει τα μέσα χρηματοδότησης με τα αποτελέσματα. Επίσης, το ΕΚΟ είναι ο δεύτερος δωρητής παγκοσμίως από απόψε πόρων Διαραστηριοποιείται παγκοσμίω, οπότε έχει πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στην ενσωμάτωση, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και ούτω καθεξής. Επίσης, έχει και πάρα πολλούς ε, επιτόπου εμπειρογνώματος εμπειρογνώμονες, εμείς ως εταίροι μπορούμε να αναζητήσουμε λύσεις για επιχειρησιακά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Είναι λοιπόν ένας πραγματικός και ανοιχτός διάλογος και μια εταιρική προσέγγιση η οποία συνήθως δεν ακολουθείται. Και εδώ στις Βρυξέλλες και επί τόπου μέσω ενός watch group που παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ μοναδικό και πολύ χρήσιμο. Και τέλος, το ανθρωπιστικό μέσο είναι πιο ευέλικτο από άλλα μέσα γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε μεταβαλλόμενες συνθήκες των κρίσεων και να προσαρμόζουμε αναλόγως το πρόγραμμα. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί όλοι θελήσαμε να διατηρηθούν εξαιρέσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια στον ε, ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Αυτό της ευελιξίας είναι ένα ζήτημα ε, για το οποίο θέτει ερωτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, όπως επίσης ε, θέτει και σημαντικούς περιορισμούς. Χρειαζόμαστε ευελιξία για τις επιχειρήσεις, ευελιξία να φτάσουμε στον κόσμο επιτόπου, να ε, μπορέσουμε να φτάσουμε σε πληθυσμούς που έχουν ανάγκη. Αυτό που δεν υποστηρίζουμε είναι ευελιξία για τις μεταβαλλόμενες προ, ε, ε, προ, πολιτικές προτεραιότητες από πλευράς Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναρωτιέται συνεχώς ευελιξία γιατί και για ποιον. Μετά από όλα αυτά, ε, εντάξει, προφανώς υπάρχουν και κάποια ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι όλα ρόδινα. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εστίαση ε, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της ε, Τουρκίας ε, που παίρνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση και αυτό εις βάρος των άλλων περιοχών του κόσμου που το χρειάζονται. Ειδικότερα φορές των κρατών μελών για την Τουρκία, κάτι το οποίο δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ της περιοχής αυτής και της Αφρικής, όπου επίσης σημειώνονται σημαντικές ανάγκες. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν εμείς, γιατί με τη βάση αυτή έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται όλοι κατά πόσο ο ΕΚΟ εξακολουθεί να λειτουργεί βάση αναγκών. Ζητούμε μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης του ΕΚΟ να αφιερωθεί σε ξεχασμένες κρίσεις. Γιατί υπάρχει μικρότερη πιθανότητα τα κράτη-μέλη να καλύψουν αυτές τις πιο ξεχασμένες κρίσεις και υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με το να συμμετέχει ο ΕΚΟ στις ε, συγκεκριμένες ε, κρίσεις. Όσον αφορά τις παρατεταμένες κρίσεις, χρειαζόμαστε ε, και επιπλέον χρηματοδότηση. 20% της χρηματοδότησης του ΕΚΟ δαπανάται σε ετήσια βάση, πρέπει όμως να συμφωνήσουμε πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι δεσμεύσεις. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι να υπάρχει για τις παρατεταμένες κρίσεις, να υπάρχει ένας τριετής προγραμματισμός με ετήσια χρηματοδότηση και προσαρμογές αν αλλάξει η κατάσταση. Ε, πάρα πολλοί άλλοι δωρητές το κάνουν αυτό, άρα μπορεί να γίνει και εδώ. Επίσης, ε, υπάρχει πάρα πολύ εστίαση στην αποτελεσματικότητα του δωρητή, δηλαδή προγραμματισμός βάσει των αποτελεσμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αποτελεσματικά, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες, κανείς δεν διαφωνεί με αυτό και η λογοδοσία είναι σημαντική, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση ότι τα λεφτά των φορολογουμένων ε, πρέπει να δαπανούνται σωστά, όμως αυτό δεν έχει προτεραιότητα σε σχέση με το τι είναι απαραίτητο για τον πληθυσμό, ε, γιατί ε, εδώ μιλάμε για την αξιοπρέπεια, τη ζωή, το θάνατο κάποιων ανθρώπων και νομίζουμε ότι στην πλάστικα χάνεται αυτή η ισορροπία. Πρέπει να βρούμε πιο εμπνευσμένου τρόπους να εφαρμόσουμε τη βοήθεια αυτή όπως κάνουν οι κάτω χώρες, ίσως μια απλοποίηση εναρμόνιση των κανόνων και των κανονισμών που ισχύουν για τους ανθρωπιστικούς εταίρους και κάτι ακόμη που τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να το κάνουν πολλές φορές και μάλιστα ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό δίνεται μεγάλη η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι ακόμη είναι κατά πόσο αλλαγές στον κανονισμό χρειάζονται ή όχι. Από το 1986 υπάρχει ο ανθρωπιστικός κανονισμός, είναι ένα από τους αρχαιότερους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όμως ο μόνος λόγος να τον αλλάξουμε θα ήταν αν μπορεί να επιτύχει, αν είναι μόνο για να επιτύχει το στόχο του. Μπορεί να το κάνει, να μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε καινοτόμοι, και ε, φυσικά εμείς έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις ε, συστάσεις ε, που έγιναν στην Παγκόσμια Σύνοδο την Ανθρωπιστική για τον προγραμματισμό κυρίως του 2012 μέχρι το 2025 οπότε υποστηρίζουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την προσπάθεια του να εφαρμοστούν ε, όλα ε, όσα έχουν συμφωνηθεί, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Θέλουμε λοιπόν ο ανθρωπιστικό μέσο να διατηρηθεί και στον επόμενο προγραμματισμό ε, με έναν προπολογισμό που να ανταποκρίνεται σε ανάγκες ανθρωπιστικές. Επίσης, να ληφθεί υπόψη στις διαπραγματεύσεις ε, για το επόμενο ε, δημοσιονομικό προγραμματισμό και επίσης κατά τη διαβούλευση στις επόμενες συμφωνίες πλαίσιο μεταξύ ΕΚΟ και μη κυβερνητικών οργανισμών να ληφθεί υπόψη ε, ε, η, αυτός ο στόχος ε, της, ε, των ανθρωπιστικών αναγκών και να τεθούν επίσης σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκερέρο ράρει το λόγο και μετά ο κύριος Γκερέρο θέλει να θέσει μια σύντομη ερώτηση. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι όμως γιατί μετά έχουμε τους καλεσμένους μας για να μιλήσουν για τη Λιβύη. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση για την έκθεση. Θα επανέλθουμε μόλις θα έχουμε και το σχέδιο έκθεσης του Ρίγκε και θα έχουμε και τις απόψεις των κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μακρογαρίσουμε πολύ τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Πριν ε, αναπτύξω την παρέμβασή μου, ε, θα ήθελα να λάβουμε υπόψη τρεις βασικές ε, σκέψεις. Πρώτον, ότι όπως λέει η μερίσια διάταξη, η συζήτηση αυτή γίνεται χωρίς έγγραφο, διότι εδώ και λίγο καιρό αποφάσισε η Επιτροπή Ανάπτυξης να κάνει μια έκθεση για την εφαρμογή αυτών των τριών μέσων και γιατί είναι και πολύ μικρότερο το διάστημα ε, στο οποίο ανέλαβα την ε, εκπόνηση της συγκεκριμένη έκθεση. Δεύτερον, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπε ο κύριος ε, Μονσερβίση. του χρόνου το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε αυτό το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο τα διάφορα μέσα και επομένως, ε, ε, από τη στιγμή που θα το παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υπάρχει μεγάλος χρόνος εντός του οποίου η Επιτροπή Ανάπτυξης θα μπορεί να εκφράσει την άποψή της για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι στην καλύτερη των περιπτώσεων η έγκριση του πολιτές δημοσιονομικού ε, πλαισίου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, επαναλαμβάνω, θα γίνει, όπως είπε ο κύριος Μονσερβίση, ταυτόχρονα με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή άνοιξη του 2019. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν η τελική έγκριση του πολιετής δημοσιονομικού πλαισίου θα γίνει με το νέο κοινοβούλιο, στη νέα θητεία. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα υπάρξει πολύς χρόνος για να μπορέσουμε να προβληματιστούμε και να λάβουμε θέση για το μέλλον. Το τρίτο ε, στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η έκθεση αυτή, ε, όπως λέει και το όνομά της, είναι ε, έκθεση εφαρμογής, δηλαδή έκθεση που εξετάζει την εφαρμογή, την εκτέλεση των στόχων και των προτεραιοτήτων, των προτάσεων που εξετάζονται στα διάφορα μέσα όταν εγκρίθηκαν αυτά τα μέσα. Και Βάσει και των κανόνων του Κοινοβουλίου, αυτή η αξιολόγηση για την Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να γίνει μέσω μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας. Και ε, χρησιμοποιώντας και ε, τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, πρέπει να σας πω ότι πρακτικά όλες οι εκθέσεις εφαρμογής που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν γίνει για νομοθετικές προτάσεις και το πώς έγινε η μεταφορά τους στις διάφορες χώρες και πώς ε, εφαρμόστηκαν στις διάφορες χώρες οι νομοθετικές υποχρεώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δει κανείς τι συνέβη στη θητεία 2009-2014, εγκρίθηκαν 23 εκθέσεις εφαρμογής όλες αυτές οι εκθέσεις ε, έπρεπε να έχουν ε, νομοθετική εστίαση και καμία δεν είχε σχέση με την Επιτροπή Ανάπτυξης ούτε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που σημαίνει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε τέτοια δουλειά ως Επιτροπή. Το πρώτο λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει βάσει στοιχείων, βάσει γεγονότων, βάσει στατιστικών στοιχείων, βάσει δεδομένων τα οποία θα μας επιτρέψουν να δούμε μέχρι ποιου σημείου πληρούνται οι προτεραιότητες, οι στόχοι, οι δείκτες και τα κριτήρια τα οποία εγκρίθηκαν όταν ε, εγκρίθηκαν τα συγκεκριμένα μέσα. Και αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τρία στοιχεία. Πώς λειτουργήσε, ποιες ήταν ε, οι ε, αδυναμίες και ποια τα δυνατά στοιχεία, τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την αξιολόγηση, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε προτάσεις για το μέλλον και πώς μπορούμε να καταφέρουμε στο μέλλον από αυτά τα διδάγματα να μάθουμε κάτι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους βασικούς μας στόχους. Σε αυτή την Επιτροπή υπάρχει πρόβλημα προθεσμιών και θα ήθελα να πω σε όλους τους σκιώδεις συγητές και εν γέννη σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, σε ποιο χρονικό πλαίσιο κινούμαστε. Θα μπορούσαμε να είχαμε γκρίνει την απόφαση για την εκπόνηση της έκθεσης μετά την παρουσίαση της πρότασης το Μάιο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα ήταν καλή απόφαση αυτή βέβαια, διότι από την έκθεσή μας πρέπει να αντλήσουμε και κάποια διδάγματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στην πρόταση της Επιτροπής και θα ληφθούν υπόψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την παρουσίαση της ε, ε, ανακοίνωση στο Μάιο. Και επίση δεν θα ήταν καλή απόφαση, διότι και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα έχει έκθεση πρωτοβουλίε και θα ήταν παράλογο αυτή να εκπονήσουν την έκθεση πριν από την παρουσίαση των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική μα πρόταση να έρθει μετά. Επομένω, πρέπει η έκθεση να έχει γίνει πριν από το Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τη θέση της τον Απρίλιο το αργότερο και α, επίσης προϋποθέτει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένο τέλη Ιανουαρίου να σας παρουσιάσω ένα έγγραφο το οποίο θα μπορεί να μεταφραστεί και στις διάφορες γλώσσες. Γι' αυτό ακριβώ ζήτησα από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας δώσει αξιολογήσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Για παράδειγμα αυτές τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Μονσερβίση και ένα συγκεκριμένο αίτημα για το ανθρωπιστικό μέσο, για το μηχανισμό αυτό, για τον οποίο ακόμα δεν υπάρχει αξιολόγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε θα λάβουμε όμως υπόψη και έγγραφα και θέσει όπως για παράδειγμα αυτά τα οποία μόλις ακούστηκαν ε, και από την Concord και από τη Voice. Άρα, συνοπτικά, πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση, να δούμε πώς λειτουργήσαν αυτά τα τρία μέσα, μέχρι ποιου σημείου είχαν κάποια προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι ποιου σημείου η πολιτική συνεργασία ήταν αποτελεσματική, αποδοτική, βιώσιμη, μέχρι ποιου σημείου η ανθρωπιστική βοήθεια δόθηκε βάση του μηχανισμού και τι αντίκτυπο είχαν στο μηχανισμό οι κρίσεις ε, που είχαμε σε ανθρωπιστικό επίπεδο για την αξιολόγηση αυτή επίση πρέπει να γίνουν, πιστεύω, και νομίζω ότι αυτό είναι και στην ε, διάθεσή μας, όχι μόνο για μένα, να γίνουν κάποιες γενικές προτάσεις, επιμένω στο γενικές, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να τις λάβει υπόψη της πριν μας παρουσιάσει την ανακοίνωσή της ε, για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει, και ακούστηκε αυτό αρκετές φορές ε, για κάποιες αυτές τις γενικές συνδέες, ε, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Επομένως, απλώς θα επαναλάβουμε αυτά ε, επί των οποίων είμαστε σύμφωνοι επί του θέματος αυτό. Επαναλαμβάνω επίσης ότι μας πιέζει ε, το χρονοδιάγραμμα γιατί πρέπει να έχουμε έκθεση πριν από το Μάιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να εκφράσει την άποψή της μετά το Μάιο, διότι η διαπραγμάτευση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα γίνει το πολύ για ένα χρόνο και επομένως ε, θα έχουμε αρκετό χρόνο να εκφράσουμε την άποψή μας. Επομένως ε, δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται όλες μας οι θέσεις σε αυτή την έκθεση, παρά το γεγονός ότι οι γενικές ε, ε, θέσεις μας και τα βασικά στοιχεία και να έχουμε τα βασικά στοιχεία για την πολιτική συνεργασία και την ανθρωπιστική πολιτική ε, στα πλαίσια της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά για τα επόμενα 7 χρόνια είναι σημαντικό να υπάρχουν. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ θα ξαναδούμε τα μελλοντικά προγράμματα όταν θα τα έχουμε. Αλλά έχεις δει ο Καλό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επηρεάσουμε τον προγραμματισμό ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Σοφχάους, θέλετε να πάρετε το λόγο, αλλά επειδή πρέπει να μιλήσουμε και για τη Λιβύη και έχουμε έναν ειδικό απεσταλμένο που θα έρθει να μας δει, έχετε μία κατεπίγουσα ερώτηση ή μπορεί να περιμένει η ερώτησή σας. Ναι, πολύ σύντομα. Σε σχέση με αυτά που άκουσα, εμένα μου αρέσουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά να σα πω την αλήθεια, προβληματίζομαι κιόλα. Κατα... Μ' αρέσουν, τη συμπαθώ, γιατί θεωρώ ότι η αναπτυξιακή συνεργασία περνάει και από τους μη κυβερνητικές, ε, τις μη οργανώσεις ε, και έχουμε συνεργασία με εσά εδώ και 25 χρόνια. Αλλά σε σχέση με την ανιχνεσιμότητα και τη διαφάνεια, ε, κοιτάξτε, αλλά τώρα για την πολιτική τώρα της διάστασης του φύλου και την αποτελεσματικότητα και για τη διακυβέρνηση, εγώ θέλω να είμαστε διαφανείς και να έχουμε και ανευνευσιμότητα, γιατί για το κράτος δικαίου όλα τα προγράμματα τα έχω δει. Έχω δει δίκαιο χωρίς κράτος, δεν υπάρχει οργάνωση και όσον αφορά το φίλο κοιτάξτε, εγώ ήμουν με ένα στρατηγό, πολύ σύντομο θα είμαι, με ένα στρατηγό όταν ήμουν στην, Αφρία, στην Αφρική, ε, μισοί στρατιώτες ήταν άντρες, μισές γυναίκες, χωρίς ε, ε όπλα ε, και ήταν μάλιστα ο Άντε εκεί ο οποίος ε, κατά τη γνώμη μου είναι εγκληματία πολέμου και ο οποίος ήταν υπεύθυνο για την ασφάλειά μας ε, με ασυρμάτους και τα πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλες, όλα αυτά τα συστήματα που σκοπό έχουν να καταστρέψουν το κράτος πρέπει κάπως να τα αντιμετωπίσουμε. Χωρίς κράτος δεν υπάρχει ανα, ανάπτυξη. Σας το λέω αυτό. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μερικές φορέ αντικαθιστούν το κράτος. Κοιτάξτε, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Δεν θα υπάρχει ποτέ αναπτυξιακή ικανότητα αν δεν υπάρχει κράτος που είναι θεμελιώδο στην, στην Αφρική και πρέπει οπωσδήποτε να το αποκαταστήσουμε. Εντάξει. Έχω εδώ τα ονόματα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ και ΔΕΦΚΟ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, ένα λεπτό έκαστος αν είναι πήγον. Μόνο αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε. Ένα λεπτό το πολύ. Όχι ολόκληρη δήλωση. Ο κύριος Κορντέρο από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτό το η φάση. Ε, ναι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ε, όπως ανέφερε και ε, ο Γενικός Διευθυντής, ο αντίκτυπος της εφαρμογής στην στον επερχόμενο προγραμματισμό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να, ακούσουμε, να δούμε τη συμβολή στις ανοιχτές διαπραγματεύσεις όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έγινε αξιολόγηση του μέσου. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη της χρονιάς ε, και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και για το Μέσο Αναπτυξιακής ε, ε, Συνεργασίας και το έγγραφο προσωπικού. Όλα αυτά θα τα λάβετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί θα μας βοηθήσουν, λέει η Πρόεδρος, στην έκθεση. Kim Ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ πάρα πολύ σύντομα όσον αφορά την πλευρά της ανθρωπιστικής βοήθειας να αναφέρω απλώς ο... Ε, και επειδή άκουσα και τα σχόλια του κυρίου Γκερέρου Σαλόμ όσον αφορά την έκθεση και τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριλάβουν να υπάρχει μια περιεκτική προσέγγιση ε, της ε, ανθρωπιστικής πλευράς είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει, υπάρχει μια έκθεση αυτή τη στιγμή ε, τελειοποιείται. Ελπίζουμε μέχρι τον Ιανουάριο να την έχετε για να μπορέσετε να τη συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας, την οποία υποστηρίζουμε και αναμένουμε βέβαια κατά τους ερχόμενους μήνες διάλογο μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν σύντομος αλλά και για τον ε, διάλογο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ε, θα υπάρξει διάλογος και στο μέλλον, ούτως ή άλλως για, τα επόμενα 18, για τους επόμενους 18, μήνες θα εξακολουθήσουμε να συζητούμε αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον και φλέγον. Κλείνουμε τώρα το σημείο 8 της ημερήσης διάταξης. Σας ευχαριστώ. Okay, colleagues, we're going to move now to... Συνάδελφοι, να περάσουμε στο σημείο 9, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, οι ανθρωπιστικές συνθήκες στη Λιβύη πάρα πολύ συζητήθηκε στο Αμπιτζάν την περασμένη εβδομάδα στην ε, Σύνοδο για την Αφρική. Μερικοί από εμά ε, ήταν παρόντε. Είναι εδώ ο κύριο Κοστέλ, ο οποίο είναι ο ειδικό επεσταλμένο τη ΥΠΑ του ΟΗΕ για του πρόσφυγε για τη διαδρομή τη κεντρική ε, Μεσογείου. Ε, ήρθαμε σε επαφή με νέου ανθρώπου που είχαν επαναπαυριστεί από τη Λιβύη στο... στην ακτή Ελεφαντοστού και είχαν τρομερέ ιστορίε να μα πούν για την εμπειρία τους στη Λιβύη, που έφτασαν δηλαδή στη Λιβύη και έπρεπε να επαναπατριστούν μετά. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε παρόν εδώ σήμερα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ανησυχούμε να ακούσουμε. Είδαμε κάποιες ε, αναφορές στο CNN και στο BBC για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας ανησυχούν πάρα πολύ Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε την κατάσταση στη Λιβύη. Ακούσαμε και δήλωση μάλιστα για την αυξανόμενη παρέμβαση του ΟΗΕ η οποία δεν έχει κάνει τίποτα για να μειώσει το επίπεδο των ε, ε, παραβιάσεων που υφίστανται οι μετανάστες. Με πολύ χαρά λοιπόν σας καλωσορίζουμε σήμερα και περιμένουμε εναγωνίως να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ε, δεν είναι δυνατόν σε μία μικρή παρέμβαση να καλύψω όλες τις πτυχές ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λιβύη, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας ε, με, για την πρόσκληση, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω κάποια πράγματα και επίσης να σας, να σας, ευχαριστήσω για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Στη Λιβύη υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες. Υπάρχει μία στατιστική που πάντοτε πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Ε, δεν σημαίνει ότι ποιο πάει στη Λιβύη θέλει να πάει στην Ευρώπη. 64%, 64 των ανθρώπων που φτάνουν στη Λιβύη έχουν φτάσει στον τελικό τους προορισμό. Σας το λέω αυτό να το θυμάστε. Η Λιβύη έχει προσελκύσει πάντοτε πολύ καιρό ε, ε κόσμο που ε, θα ήθελε να παραμείνει στη Λιβύη. Πόσοι είναι οι αλλοδαποί δεν ξέρουμε. 700.000 λέει η Αφρικανική Ένωση, άλλοι λένε ένα εκατομμύριο, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστων ε, λέει περίπου 300.000, ε, τώρα για τους ε, πρόσφυγες, 43.000 ε, είναι οι πρόσφυγες, κυρίως από το Συρία, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, και κάποιους Σομαλούς και Ερυθρέους από την Ανατολική Αφρική και κάποιοι Σουδανοί. Είναι σημαντικό να πούμε ε, ότι ε, η Λιβύη ποτέ δεν έχει εγκρίνει τη σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες, αλλά την σύμβαση για τους πρόσφυγες του 1969 ισχυρίζεται όμως ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και απορρίπτει την ιδέα ότι έχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από τη σύμβαση αυτή. Ε, σήμερα έχουμε δύο δύσκολε καταστάσει. Να μην ξεχνάμε του Λίβιου. Υπάρχουν και οι Λίβοι οι οποίοι επηρεάζονται από την σύγκρουση. Περίπου μισό εκατομμύριο που έχουν εκτοπιστεί λόγω της ε, ε, σύγκρουση, χρειάζονται την υποστήριξή μας και πρέπει να τους βοηθήσουμε δήμου δήμους οποίους βρίσκονται, ε, που έχουν εκτοπιστεί δηλαδή, για να μπορέσουν να επιστρέψουν στον τρόπο της προηγούμενη κατοικία τους, προηγούμενη πριν από τη σύγκρουση. Τώρα, για τους 43.000 πρόσφυγες που ζουν ε, εκτός ε, των κέντρων κράτησης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 2.000 πρόσφυγες στα 30 κέντρα κράτησης τα οποία διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα κέντρα κράτησης στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση ε, και τα οποία διαχειρίζονται διάφορες ε, παραστερωτικές οργανώσεις και διάφοροι λαθρέμποροι. Ε, αυτά τα κέντρα κράτησης ε, και η κυβέρνηση τα ελέγχει, ε, αλλά υπάρχουν και άλλα κέντρα κράτησης τα οποία ελέγχει η κυβέρνηση σε άλλα σημεία της Λιβύης. Δεν ξέρουμε πόσα είναι. Θα ήθελα επίσης να μην ξεχνούμε ότι μεταξύ όσων πηγαίνουν στη Λιβύη υπάρχουν και οι οποίοι πηγαίνουν μετά στην Ευρώπη, επειδή συχνά υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι είναι όλοι οικονομικοί μετανάστες. 74%, 74% των ανθρώπων που από την Ανατολική Ευρώπη πηγαίνουν στη Λιβύη και μετά πηγαίνουν στην Ευρώπη, παίρνουν κάποιο είδους προστασία στην Ευρώπη. Όταν αφορά τώρα τις, τις διόδους της Δυτικής Αφρικής, 24%. 24%. Δεν είναι λοιπόν όλοι οικονομικοί μετανάστες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από πολεμικές συγκρούσεις ή από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους. Εμεί επιχειρούμε υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκε στη Λιβύη, μερικές φορές μας κατηγορούν. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά μα κατακρίνει για την υποστήριξη της κυβέρνησης της Εθνικής ε, Ομόνιας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ε, οι συνθήκε. Ε, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε ζωέ. Σα το λέω, έχουμε και εμεί ηθικά διλήμματα όταν πηγαίνουμε σε κέντρα κράτηση στη Λιβύη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχά, ε, έχετε γύρω σα ε, του σωματοφύλακέ σα, έχετε πάρα πολλού αξιωματούχου ε, τη Λιβύη. Δεν μπορεί να έχετε εμπιστευτικέ συζητήσει με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν κάνει κανεί τη λάθο ερώτηση, ε, υπάρχει περίπτωση αντιπίνων. Δεν ξέρετε ότι θα μπορέσετε την επόμενη μέρα να ξαναπάτε στο κέντρο κράτη. Μερικέ φορέ θέλουμε να αποσυρθούμε, θέλουμε να φύγουμε, αλλά μα λένε σα παρακαλούμε, ελάτε, γιατί είστε μάρτυρες ε, του πόσο υποφέρουμε. Ε, δηλαδή τα λίγα που ε, μας, μας, δίνεται είναι καλύτερα από το τίποτα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρεί κανείς υπό αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και φυσικά έχουμε ηθικά διλήμματα. Είναι δύσκολο Κάνουμε, υπάρχει κάποια πρόοδος ε, με την κυβέρνηση, έχουν δεχθεί την ε, περασμένη εβδομάδα ε, να δημιουργήσουν ένα κέντρο στην Τρίπολη όπου θα μπορούν να υποδέχονται άτομα που απελευθερώνονται από τα κέντρα κράτηση με κάποια εμπιστευτικότητα, κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις προσφέρουν τη βασική υποστήριξη πριν να φύγουν. Η μόνη χώρα που έχει αποδεχθεί την εκένωση είναι ο Νίγηρας. Ε, ο Νίγηρας δεν είναι όμως Λιβύη, είναι πρόσφυγες στη Λιβύη, έτσι. Έχουμε κενώσει μια μικρή ομάδα την περασμένη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε ε, στις 12 και στις 19 Δεκεμβρίου. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις με διαφορετικούς ανθρώπους για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τις φυλακές και να φύγουν και από τη Λιβύη. Οπότε έχουμε σημειώσει τη, τα συμπεράσματα ε, της ε, Συνόδου ε, στο Αμπιτζάν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε την εκένωση των προσφύγων από τη Λιβύη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι από πλευράς προσφύγων έχουμε τον περιορισμό των 7 ηθαγενειών. Ιράκ, Συρία, Παλαιστίνη, Σομαλία, Ερυθρέα, Αιθιοπία, και Σουδάν ανέρχονται από τον Ταρβούρ. Άλλοι πρόσφυγες όπως κεντροαφρικανικής δημοκρατίας, ε, Μάλι, ε, κάποιοι που φεύγουν για να διαφύγουν του Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Προσπαθούμε λοιπόν, έχουμε ένα μηχανισμό ε, αναγνώρισης. Δεν θέλουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στις χώρες τους ε, όπου θα εκτοπιστούν ή που θα έχουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ή θα παραβιαστούν τα τρόπινα δικαιώματά τους. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η έκκληση να φύγουν οι πρόσφυγες από τη Λιβύη δεν θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου επιστροφή θα είναι η μόνη λύση καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και άλλες χώρες της διεθνούς κοινότητας να επιδείξουν αλληλεγγύη σε σχέση με τον Ήγηρα, γιατί η εκένωση στον Ιγυρία ε, δουλεύει μόνο αν υπάρχει αλληλεγγύη με τον Ήγηρα. Επομένως δεν θα πρέπει να μείνει ο κόσμος εκεί για πάντα. Ε, έχουμε πει στις αρχές του Νίγηρα ότι θα μετεγκαταστήσουμε τους περισσότερους που θα φύγουν από τη Λιβύη για να πάνε στον Ήγηρα. Δεν έχουμε δει πολλή αλληλεγγύη με την Ιταλία, μόνο οικονομική αλληλεγγύη. Ελπίζουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη με τον Ήγηρα ως προς τις υποσχέσεις μετεγκατάσταση, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Ένα από τα, από τις, μία από τι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, όπως ε, ακούσατε υπάρχουν δυσκολίες ε, με τη διάσωση στη θάλασσα, ο κόσμος αποβιβάζεται σε διάφορα σημεία στις ακτές, σε 12 σημεία στις ακτές της Λιβύης. Προσπαθούμε με τον ΟΗΕ να τους βοηθήσουμε πριν να πάνε ε, στον, ε, ε, στα κέντρα κράτησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την κατάσταση μιας μεμονωμένης περίπτωσης που είδαμε για μερικά λεπτά ή για μερικές ώρες σε αυτά τα σημεία αποβίβασης. μετά από λίγο καιρό μάλιστα επιστρέφουν στις Ιταλικές ακτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει από τα κέντρα κράτησης στα, στα οποία πήγαν ε, ο Γενικός Γραμματέας είχε πει ε, στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις, ε, της, των αρχών της Λιβύης που συνεργάζονται με τους λαθρεμπόρους. Άρα πολύ περισσότερο πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι το σχέδιο της Αφρικανικής Ένωσης είναι να αδειάσει τα κέντρα κράτηση ε, στη Λιβύη, αλλά ας μην έχουμε αυταπάθε. Κάθε φορά που φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, ε, μετά ε, γεμίζουν με άλλους την επόμενη μέρα. Οπότε ας μην ξεχνούμε το βασικό μας στόχο. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση και την ε, εξαγρίωση που ακούστηκε, ε, που έδειξαν αυτές, αυτά τα δελτία του CNN και του BBC για την εκμετάλλευση των μεταναστών και των ε, προσφύγων στη Λιβύη. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι το καινούριο. Καταρχάς δεν αφορά μόνο τη Λιβύη. Αυτές τις ιστορίες τις ακούμε από την πτώση του καθεστώτος του Καντάφη όταν πήγε ο κόσμος στο σύνορο με την Αίγυπτο και με την Τινησία. Δυστυχώ δεν είναι κάτι το καινούριο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διασώσουμε περισσότερο κόσμο σε άλλε περιοχές όπου δεν έχουμε πρόσβαση. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, να σα πω την αλήθεια. Ελπίζουμε όμως ότι η διεθνής κοινότητα θα βοηθήσει, την, θα υποστηρίξει την αναθεώρηση του ειρηνευτικού προγράμματος της Λιβύης για να δούμε τι εισρωή θα υπάρξει ε, ε, και να υπάρχει και κράτος δικαίου γιατί διαφορετικά θα υπάρχει ατιμορρησία για τους λαθρεμπόρους, μερικοί είναι πάρα πολύ γνωστοί και όσο υπάρχει ατιμορρησία το λαθρεμπόριο ανθρώπων θα συνεχίσει για το άμεσο μέλλον. Θα σταματήσω εδώ. Αν έχετε ερωτήσει, ευχαρίστω να τι ακούσω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τι ερωτήσει, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είπατε ότι όσον αφορά τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ε, ποιος τελικά ασχολείται, γιατί υπάρχουν διάφοροι που ασχολούνται και όταν είπατε για υποσχέσεις εγκατάστασης στο Νίγηρα, εννοείται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα δέχονται αυτούς που έχουν περάσει από αυτά τα κέντρα. Δηλαδή, ε, σε αυτή τη συμφωνία καταλήξατε στο Αμπιτζάν. θα είχα να ρωτήσω. Λοιπόν, όσον αφορά τον Διεθνή Οργανισμό ε, Μετανάστευσης, αυτοί εξακολουθούν να ασχολούνται με εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν στον Ήγηρα ή κοιοθελώς. Η και ο θελός. η κορυφής στο Αμπιτζάν απλά ε, αναφέρει και επιβεβαιώνει ότι όσοι θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μπορούν να το πράξουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν τελικά αυτό το ντοκιμαντέρ του CNN ίσως ε, να τρακούνησε τη συνείδηση κάποιων κρατών της ε, Αφρικής. Ίσως και ελπίζουμε και να είναι το βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Η πατερμοστία προσφύγων ασχολείται μόνο με εκείνους που έχουν χαρακτηριστεί πρόσφυγες. Αλλά η κυβέρνηση της Εθνικής Ομόνοιας της Λιβύης δεν θέλει αυτή να πηγαίνουν απευθείας ε, από τη Λιβύη σε άλλες χώρες όπου θα έχουν αγροσίες πρόσφυγες γιατί φοβούνται ότι θα μαζευτούν τελικά όλοι στη Λιβύη. Ε, θα μπορούσαν και από τον Ήγυρα να πάνε σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καναδά και αλλού και άλλοι έχουν δεχτεί ε, να δέχονται πρόσφυγες από τον Ήγηρα. Τώρα, γκρίζε ζώνη είναι εκείνες οι εθνικότητες που προς το παρόν δεν έχουν ε, γίνει δεκτές. Κάποιοι, ας από το Μαλί δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Μαλί. Δεν θέλουμε, λοιπόν, αυτοί να μπουν σε αυτό το μηχανισμό επαναπατρισμού χωρίς να είναι σαφές από πού προέρχονται, γιατί εγκατέλειψαν τη χώρα. Θέλουμε να έχουμε και διαφοροποιημένες, διάφορες λύσεις. Να ξέρουμε πρώτα απ' όλα γιατί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και ξεκινάμε τις ε, ερωτήσεις. Νομίζω ότι κάποιοι ε, οικειοθελώς επιστρέφουν, αλλά άλλοι πάλι όχι ε, οικειοθελώς ο κύριος Κεραίρο και μετά έχω ένα μακρύ κατάλογο που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν και επιπλέον διότι πολλά από αυτά τα οποία ήθελα να ρωτήσω τα απαντήσατε απευθεία στην παρέμβασή σας. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση σε ανθρωπιστικές κρίσεις, ε, συνήθως έχουμε πολύ ε, καλά καθορισμένο και σαφές τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και πολλές φορές ε, οι κρίσεις αυτές είναι ανθρωπιστικές κρίσεις και από κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται και προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι η περίπτωση της Λιβύης. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο γενναιοδορή και ε, βοηθά λιγότερο τελικά στην επίλυση των προβλημάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη στην πραγματικότητα με την πρόταση που ε, προέκυψε στο Αμπιτζάν όπου κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, θα ε, διέθεταν αεροπορικά μέσα για τη μεταφορά περίπου χιλίων ατόμων που πολλούνταν ως ε, σκλάβοι στη Λιβύη και κατά πόσον υπάρχουν ε, και κάποιες διευκολύνσεις για τα παιδιά των ε, προσφύγων, εάν υπάρχει δυνατότητα για σχολική εκπαίδευση κάπου στη Λιβύη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε. Κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή ότι συμμερίζομαι πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Κοστέλ, κυρίως αυτά τα οποία είπατε σχετικά με το ντοκιμαντέρ αυτό που προέβαλε το CNN και ότι τελικά δεν είναι και κάτι το καινούριο, όλοι το ξέραν έχουμε μία έκθεση του περασμένου Δεκεμβρίου όπου η Λιβύη αναφέρεται και χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλής χώρα. Και τον Απρίλιο αυτού του έτους ε, έχουμε και μια έκθεση του ΙΕ νομίζω που λέει ότι πολλούνται οι ε, μετανάστες ως σκλάβοι. Ερωτώ λοιπόν τώρα, η Λιβύη είναι χώρα ασφαλής ή δεν είναι. Και άλλη μια ερώτηση που αφορά στις αποφάσεις που λήφθησαν στο Αμπιτζάν. Θα ήθελα να γνωρίζω τελικά αυτά τα ιδιαίτερα κατεπήγοντα, τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος ε, Μακρόν. Αυτό πώς θα υλοποιηθεί, με ποια μέσα, στρατιωτικά, αστυνομικά. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι Υπάρχουν κέντρα κράτησης όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και όπου κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει τίποτα. Σχετικά με τους επαναπατρισμούς, θα ήθελα να γνωρίζω το εξής. Είναι κάτι που με ανισχύει πάρα πολύ. Τι διαδικασίες ακολουθούνται, ποιες είναι οι Ο πρόεδρος Μακρόν είπε σε συνέντευξή του στο Αμπιτζάν ότι αυτοί οι παναπατρισμοί είναι οικειοθελείς. Και την προηγούμενη μέρα η Μπουρκίνα Φάσο μίλησε για μία δράση επαναπατρισμού, χωρίς όμως να αναφέρει ότι θα είναι οικειοθελείς αυτή οι επαναπατρισμή, μπορεί να είναι και εξαναγκαστική. Ε, θα ήθελα λοιπόν επ' αυτού να έχω και τη δική σας την άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη ήταν επιτόπου και συναντήθηκε και με συγκεκριμένου ανθρώπου. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε και κύριε Κοσετέλ, να πάμε ε, λίγο σε αυτή τη συμφωνία που αναφέρεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του IMO, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, διάφορων οργανισμών, το αναφέρατε. Αλλά θα ήθελα να έχω μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πώς γίνεται ο έλεγχος αυτών των ανθρώπων. Γιατί λέγεται ότι πριν από τα Χριστούγεννα περίπου 15.000 άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν στη Λιβύη. Και από ό,τι έχω καταλάβει ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει ε, πρόσβαση ε, στις πρεσβείες, αλλά το να απευθυνθεί κανείς στις πρεσβείες για να μάθει πληροφορίες για τους πολίτες τους είναι πολύ πιο δύσκολο. Υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, γιατί δεν είναι απαραίτητα Σύριοι και Παλαιστίνοι. Ε, μπορεί να είναι και ε, Σουδανοί και άλλοι, όποιο να είναι. Υπάρχει ε, λοιπόν κάποιος εσωτερικό έλεγχος για να είναι σαφές ότι πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες. Θα ήθελα να μα ενημερώσετε από αυτού. Και κάτι άλλο. Εσείς ε, μιλήσατε για αυτά τα κέντρα κράτησης που είναι εκτός ελέγχου, δεν ελέγχονται από το κράτος. Πήγαμε πριν από λίγα και λίγους μήνες ε, στην ε, Τρίπολη και εκεί είχαμε την εντύπωση ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε αυτά τα κέντρα κράτησης και δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε κρατικά και μη κρατικά κέντρα κράτησης. Εσείς έχετε τέτοιου πληροφορίες και αυτά τα μη κρατικά κέντρα υπάρχει δυνατότητα να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά. Αυτά προς το παρόν. Η κυρία Κέγγε, που και αυτή ήταν, ήταν παρούσα στο Αμπιτζάν. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Εμείς ε, συναντηθήκαμε με τους ανθρώπους ε, ε, που επιστρέφουν ε, στη Λιβύη. Εγώ διάλεξα όμως κάτι άλλο. Ξέρετε τι έκανα. Εγώ πήγα στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, το μεγαλύτερο οικονομικό τετράγωνο του Αμπιτζάν, όπου η ΜΚΟ ασχολούνται με αυτούς που εργάζονται στον τομέα του ξύλου και της επεξεργασίας του ξύλου. Η δυνατότητα λοιπόν να υπάρχει απασχόληση, να κάνουν οι άνθρωποι κάτι, να κατανοήσουν ότι έχουν μέλλον. Μαζί με αυτούς είδαμε και κάποιους άλλους που γύρισαν πίσω και αυτοί όμως εκεί που εργαζόντουσαν θα, κατα... αναγερθεί μία γέφυρα σας λέω λοιπόν ότι σε αυτό το μεγαλύτερο οικοδομικό τετράγωνο του Αμπιτζάνη οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε και μας ζήτησαν να ξεκινήσει η συζήτηση με την κυβέρνηση για να δούνε τελικά τι θα κάνουν, πώς θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι, να μετεγκατασταθούν και αυτό είναι επίγον γιατί η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτούς ακόμα και όταν κάνουν ε, κάποιες ε, ε, για υποδομή δεν ασχολούνται με το τι θα κάνουν ε, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί που θέλουν να χτίσουν. Ε, παραδείγματος χάρη προηγουμένως ακούσαμε για γέφυρα. Ε, άρα δηλαδή το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να εφαρμόζει μια καλή πολιτική επιτόπου να επεμβαίνει ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μετακινηθούν. Σας μιλάω για το Αμπιτζάν γιατί εκεί όλοι μας καταδικάσαμε τη δουλεία, καταδικάσαμε την λαθροδιακίνηση και θέλω να αποκαλύψω και κάτι άλλο το οποίο είπε και ο κύριος Καστέλ, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κάποια στιγμή ο κύριος Καστέλ είπε, ελπίζω ε, να μην συμβεί ότι έγινε με την Ιταλία και τον Ήγηρα. Η Ιταλία, ξέρετε, δούλεψε μόνη της ε, και επικρίθηκε όμως σε μια χρονική στιγμή όπου κανένα κράτος μάλιστα, ή μάλλον δεν θέλανε όλα τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν την Ιταλία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν τελικά δεν υπάρξει μια ολιστική διαφορετική προσέγγιση. Εάν δεν επικρατήσει πράγματι ίσης, ίσως επιμερισμός των ευθυνών, ε, τελικά θα συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος εισαγωγικά να είμαστε κρατημέλη, ποιο ε, τα κάνει καλά και ποιο όχι. Σήμερα νομίζω ότι πρέπει βεβαίω και να δείξουμε αλληλεγγύη έναντι στον Νίγηρα, αλλά γενικότερα θα πρέπει να ασχοληθούμε πώς πρέπει να επέμβουμε στην Αφρική με νόμιμους τρόπους. Γιατί Κατά την άποψή με αυτή η task force που υποτίθεται αποφασίστηκε στα Μπιτζάν, πώς θα επεμβαίνει μακροπρόθεσμα, τι θα γίνει τελικά. Θα δουλέψουμε περισσότερο για νόμιμες διόδους, να υπάρχει μεγαλύτερη μετακίνηση. Εγώ θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί έχω την εντύπωση ότι σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε, το μόνο που απασχολούσε ήταν πώς θα βιάσει η Λιβύη. Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ποια είναι τα εργαλεία ε, που θα έχει η Task Force ε, τι δυνατότητες θα έχει η Task Force, θα μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας. Εμείς ε, θέλουμε απαντήσεις, όχι μόνο ένα κράτος μέλος μόνος του, αλλά όλα μαζί. Και δεν πρέπει να δεχόμεθο ένας επιθέσει από τον άλλο, γιατί αν δεν υπάρχει ελληνική, νομίζω ότι αυτό είναι πετιότητα όλων. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερφιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοστέλ για την ειλικρίνειά του και τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσετε την παρέμβασή σας, κυρίως υπενθυμίζοντας ε, τη δύσκολη διαφορά μεταξύ οικονομικού, πρόσφυγα, ε, οικονομικού μετανάστη και πρόσφυγα. Δεν έχω τα στοιχεία τώρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που ζητούν από την Ανατολική ε, Αφρική καθεστώς ασύλου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που πρέπει να αναγνωριστούν ως οικονομικοί πρόσφυγες και πολλοί ε, θεωρούνται οικονομικοί μετανάστες. Δεν είναι απλά τα πράγματα λοιπόν ε, και ακόμα και από την ίδια την υπατερμοστία για τους πρόσφυγες οι προνομιούχοι είναι αυτοί, μάλλον αυτό το οποίο προτιμούμε είναι επιστροφή προς τις χώρες ε, καταγωγής, ε, δηλαδή προς το Σουδάν. Ε, τι κάνουμε τώρα για τα θέματα αυτά, διότι εκεί υπάρχει μια μερική συμφωνία. Και επίσης τι κάνουμε για να σεφαστούμε και αυτά τα οποία αναφέρατε για την Δυτική Αφρική το δικαίωμα του ασύλου και τη δυνατότητα του καθενό και το δικαίωμα του καθενό σε προστασία. πώ αντιμετωπίζεται αυτό στις χώρες. Ένα δεύτερο θέμα, ε, στο οποίο επίσης ήσασταν ιδιαίτερα ειλικρινείς, όπως και η Τζούντιθ και εγώ ήμουνα στην αποστολή στη Λιβύη για από την Επιτροπή Λίμπε, που πήγε και στην ε, ε, την Ισία τελικά γιατί δεν μπόρεσε να πάει στη Λιβύη και συναντήσαμε και εκπροσώπους ε, της Λιβύης ε, και ξέρω ότι ε, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ε, δίστασε να δεχτεί να προσφέρει βοήθεια για την φόρτωση στα σκάφη. Ξέρουμε ότι εκεί είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά υπάρχουν προβλήματα μπορούμε να τους βρούμε στην Ιταλία ή στη Λιβύη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή επιβιβαστούν επί ενός σκάφου, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να βρεθούν ε, τελικά ε, ελεύθεροι ή θα βρεθούν κάπου σε χώρους που θα τους πουλήσουν ως δούλους. Ε, θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις περαιτέρω λοιπόν για το θέμα αυτό. Το ίδιο όσον αφορά τα κυβερνητικά κέντρα. Τι σημαίνει κυβερνητικό κέντρο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το ερώτημα, αλλά η κυβέρνηση, ε, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τη διεθνή κοινότητα ελέγχει ένα ελάχιστο τμήμα της Λιβύης, πάρα πολύ μικρό τμήμα. Επομένως, πώς μπορεί να ε, εφαρμοστεί η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης. Ε, εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε μόνο με την Λιβική κυβέρνηση, που σημαίνει ότι η πλειοψηφία της ε, Λιβύης είναι εκτός ελέγχου. Η πλειοψηφία των προσφύγων που βρίσκονται στα κέντρα είναι εκτός ε, ελέγχου, στα χέρια παραστρατιωτικών ομάδων και φυσικά ξέρω ότι δεν μπορείτε να κάνετε θαύματα, ξέρω ότι είναι δύσκολε οι συνθήκες και ξέρω ότι υπάρχουν και δεντολογικά προβλήματα για τους εκπροσώπους της ΥΠΑ της Αρμοστίας για την πρόσφυγη για τους πρόσφυγες επιτόπους. Πέστε μας όμως λίγο πιο σαφώς πώς έχουν τα πράγματα για την πραγματική κατάσταση σε όλη τη Λιβύη και πιστεύω ότι όλες οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν πρέπει να αναλυθούν αρκετά νωρίς. Υπάρχει ε, ε, μια επιτροπή διέλευσης που θα συστηθεί στη ε, Τρίπολη, αλλά δεν ξέρουμε ε, τι θα γίνει με την ε, κυβέρνηση, τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Είναι πολύ περίπλοκη λοιπόν η κατάσταση και ακόμα και μετά από αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης δεν πρέπει να λέμε ψέματα στην κοινή γνώμη, πρέπει να τους λέμε πώς έχει στην πραγματικότητα η κατάσταση. Ε, δεν θα ρυθμιστούν τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε σχέσεις με κυβερνητικές ε, οργανώσεις ε, για την κατάσταση στην Ανατολική Λιβύη και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όπως και εσείς πιστεύω ότι μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από το αδιέξοδο, αλλά είναι και αυτή πάρα πολύ δύσκολη. Μόλις ήρθα από μια συνεδρίαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όπου συζητήθηκε το ίδιο θέμα και επίσης τελευταίο ζήτημα αυτό το οποίο βλέπω να αυξάνεται συνεχώς είναι ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης του Νίγηρα, διότι υπάρχει κάτι το οποίο βαραίνει πάρα πολύ τον Νίγηρα. Μας είπατε ότι είναι η μόνη χώρα που δέχεται επανεγκατάσταση ε, ε, από τη Λιβύη και τολμώ να πω ότι και η Τινησία έκανε κάποιες αντίστοιχες ε, προσπάθειες αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος και για τον Ήγηρα. Και εσείς πώς αναλύετε την κατάσταση στο βόρειο Ήγηρα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Είχα και κάποιες ερωτήσεις λοιπόν περί σαφήνες. Ο Χουαν Φερνάντο Λόπες, ο οποίος και αυτός ήταν στο Αμπιτζάν. Ακριβώς. Ευχαριστώ Λίντα. Ήθελα να αναφερθώ στην ίδια εμπειρία που ζήσαμε κάποιοι από εμά που συμμετείχαν εκεί στο Αμπιτζάν την περασμένη εβδομάδα, σε αυτή την ε, σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης. Ε, έχουμε ήδη τις δηλώσεις ε, που εγκρίθηκαν, αλλά αυτό το οποίο είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτές οι πρακτικές δουλείας δεν είναι καινούριες, συνεχίζονται εδώ και χρόνια. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν έρχεται ακριβώς να σταθεί σε αυτό τι καινούριο υπάρχει σε αυτή την κατάσταση ε, που έχει εξοργήσει ε, επειδή ακριβώς ε, δημοσιοποιήθηκαν οι πρακτικές που εφαρμόζονται από τους δουλεμπόρους και τους διακινητές, από ετούντες άσυλο, αλλά και από οικονομικούς μετανάστες. Τι νέο υπάρχει. Απλώς το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε. Ε, η κλίμακα του προβλήματος, το επίπεδο της ατιμορρησίας. Και όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση ενός μαζικού ανθρωπιστικού προβλήματος, ε, ένα σύστημα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τεράστια κλίμακα, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν απλώς να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες σχέσεις, σκέψεις όσον αφορά τις επιλογές που γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Ανθρωπιστικές σχέσεις, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή ε, με μετανάστες της Ποσαχάριας Αφρικής, οι οποίοι είχαν και τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην ε, ακτή του Ελεφαντοστούν και να επιστρέψουν μέσω προγραμμάτων ε, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς και από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστασης βεβαίως, αλλά υπήρχε και ε, συμμετοχή της ΥΠΑ Αυτό που ακούσαμε από αυτούς είναι ότι χρειάζεται δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της κοινωνικής και οικονομικής πρόοδου και πρέπει να βοηθήσουμε και για την επιβολή του νόμου και την καταπολέμηση της, ας τη έτσι, της εμπορικής διάστασης αυτής της αγοραπολισίας ανθρώπων. Ε, σίγουρα πρέπει να μάθουμε για αυτή την αλυσίδα για να μπορέσουμε να τη διαρρήξουμε αλλά θα μπορέσουμε να διαρρήξουμε αυτή την εμπορική κλίμακα αγοραπολισίας ανθρώπων. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει ε, μια task force η οποία πραγματικά θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τον νόμο και να σπάσει αυτή την αλυσίδα. Ε, υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε ε, να εξετάσουμε σε ενδεχόμενο. Ωραία, θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχει συμφωνηθεί. Μας ε, είπατε κάποια στοιχεία, είπατε 26% από τη Δυτική Αφρική ε, μπορούν να λάβουν καθεστώς πρόσφυγα. ο εθελοντικό επαναπροτισμός είναι ε, από τη Δυτική Αφρική που επιστρέφουν στην ακτή του ελεφαντοστούν και ούτω καθεξής. Και αυτό το νέο κέντρο επεξεργασίας ή δεν ξέρω πώς αλλιώς αποκαλείται στη Λιβύη θα είναι από χώρε της Ανατολικής Αφρικής ε, όπου ε, κατά πάσα πιθανότητα θα δεχτούν να τους δοθεί και καθεστώς πρόσφυγα. Ο Νίγηρας δεν δέχεται λοιπόν μόνο ανθρώπους από τον Ήγηρα, αλλά δέχεται να υπάρχει κάποιος καταβλισμός, ένα κέντρο στο οποίο ε, θα έχουμε εκτοπισμένα άτομα από όλη την Αφρική ή κάποιοι που εκ πρώτης αναλύσεως φαίνεται ότι μπορούν να λάβουν καθεστώς πρόσφυγα. Κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν. Τι σχεδιασμός υπάρχει γενικότερα. Υπάρχει σχεδιασμός. Ε, για να δούμε και κάποια από τα ανθρωπιστικά στοιχεία που έχουμε δει. Να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσει. Η Πατρίτσια Τόγια θέλει το λόγο. Θες να πεις δύο πράγματα. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τις ερωτήσεις για μεγαλύτερη ε, σαφήνεια όσον αφορά τη δυνατότητα να υπάρχει ένα πρόγραμμα υπό αυτές τις συνθήκες να μπορέσω να καταλάβω λίγο περισσότερο για το τι θα μπορούσε να συμβεί στο θέμα αυτό των ε, εκτοπισμών ε, για ανθρωπιστικούς λόγους από τους ε, ε, καταβλισμού ε, στη Λιβύη και συμφωνώ και με αυτά που είπε η συνάδελφος Κιέγγε που νομίζω ότι έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη παρέμβαση. Μια επιπλέον ερώτηση ε, βάσει αυτών που έλεγε προηγουμένω και η Λίντα. Μα είπατε ότι όσον αφορά την Δυτική Αφρική ένα 24% θα μπορούσε να λάβει καθεστώς πρόσφυγα, ενώ ένα 74% αν κατάλαβα καλά όσον αφορά τα άτομα που προέρχονται από την Δυτική Αφρική δεν θα μπορούσαν να λάβουν καθεστώς. Μπορείτε να μας τα δημοσιοποιήσετε σε αυτά τα στοιχεία, διότι στη χώρα μου υποστηρίζετε ότι όλοι είναι οικονομικοί μετανάστες και πρέπει να κάτσουν σπίτι τους. Και αυτές φυσικά δεν είναι και οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά και πιο... Ε, προχωρημένες ε, ε, δυνάμεις οι οποίες έκαναν ολόκληρη εκστρατεία απονομιμοποίησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων ισχυρίζονταν ότι θα μπορούν ε, πλέον να είναι και οικονομικοί μετανάστες και θα ήθελα να έχω αυτά τα στοιχεία για να τα δημοσιεύσω για να τους πω ότι δεν πρόκειται μόνο για οικονομικούς μετανάστες αλλά για ανθρώπους που έχουν άλλη τραγωδία στην πλάτη τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε και μια νομική βάση για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε ε, έστω και χωρίς συνεκτικό τρόπο, ε, μια δυνατότητα νόμιμης εισόδου. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε οδηγία για τον επαναπατρισμό, ε, ξεκινήσαμε από την ουρά. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή και τώρα και αυτή τη δυνατότητα νόμιμων εισόδων, γιατί μόνο η νομιμότητα είναι αυτή η οποία κερδίζει έναντι όλων των υπολείπων, ποια είναι η πράγματι οικονομική μετανάστες, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς και επιτρέψτε μου να σας πω ότι με εξέπληξε να διαβάσω ότι η ύπατη αρμοστία ευχαριστεί την ε, γαλλική κυβέρνηση που δέχτηκε 25 πρόσφυγες στους οποίους είχαμε εκτοπίσει από τη Λιβύη. Δηλαδή τι θα γράφαμε αν η γαλλική κυβέρνηση ή κάποια άλλη κυβέρνηση σε περίοδο μεγαλύτερης εισρωής στην Ιταλία είχε πει «Ε, για μια φορά δέχομαι να έρθει ένα σκάφος ε, το οποίο υποδέχεται και ε, σώζει ζωές ε, να έρθει σε ένα γαλλικό λιμένα ή σε έναν ισπανικό λιμένα. Αυτά είναι αλληλεγγύη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι συνεντέξει τύπου στο Αμπιτζάν για άλλα πράγματα. Αλληλεγγύη και αλληλεγγύη και πάλι. Ευχαριστούμε τη Γαλλία, αλλά όχι για να του στήσουμε και μνημείο. Thank you. There were a lot of questions. Ευχαριστώ πολύ. Πολλέ ερωτήσει υπήρξαν από του συναδέλφου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοστέλ για να απαντήσει και ξέρω ότι η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να πούν κάτι. Αλλά πρώτα να απαντηθούν οι ερωτήσει γιατί μετά μπορεί να θέλετε να προσθέσετε κάτι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω τηλεγραφικά να απαντήσω και αν θέλετε να λάβετε και άλλες ε, ε, διευκρινήσεις μπορείτε να το κάνετε μέσω του γραφείου μας στις Βρυξέλλες το κείμενο τη σύντομη δήλωση ε, από το Αμπιτζάν δεν είναι πολύ σαφέ σε σχέση με το τι θα συμβεί, οπότε έγινε μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση στην Αντίσα Μπέμπα σήμερα το απόγευμα τη Task Force και βασική εστίαση τη Task Force ε, ήταν ε, τα δικαιώματα αποβίβαση από τα αεροπλάνα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει περισσότερη πρόσβαση από τα αεροπλάνα από τις αφροκανικές χώρες στη ακριβή για να μπορέσουν να πάρουν πίσω τους πρόσφυγες και να τους πάνε πίσω στις χώρες προέλευσής τους. Δεν γίνεται τίποτε παραπάνω για την ώρα, αλλά περιμένουμε διευκρινήσεις για την κατάσταση των παιδιών και τι μπορεί να γίνει για τα παιδιά. Υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός ασυνόδευτων ε, παιδιών ε, στη Λιβύη που βρίσκονται στα κέντρα ε, κράτησης 54 από αυτά τα παιδιά θα φύγουν, ε, κάτω των 14 ετών είναι, μερικά είναι και 6 ετών, οι γονείς τους δεν ξέρουμε που είναι ή αν ε, είναι στη ζωή. Θα τους πάμε στον Ήγηρα και θα αποφασίσουμε βάσει του καλύτερου συμφέροντός τους ε, ποια είναι η καλύτερη λύση, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους γονείς τους, ε, θα κάνουμε οικογενειακή επανένωση, χώρες προέλευσης, οποιαδήποτε λύση για να μπορέσει να υπάρξει ένα μέλλον για αυτά τα παιδιά. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος ε, Μακρό, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του, δεν ξέρω τι είπε, τι δεν είπε, έγινε συζήτηση από ό,τι κατάλαβα για την αστυνομική δύναμη στο Αμπιτζάν, ε, είδα κάποια κάποιες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, ε, αλλά δεν, ε, τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία άποψη ως προς την αστυνομική ή στρατιωτική συνοδεία ή οτιδήποτε. Κάποιοι εξημών μιλήσατε για τα ε, για τους καταβλισμούς, στα στρατόπεδα. Έχουμε φρικτά κεντρικά ε, και συγγνώμη, κέντρα κράτησης, ε, είναι αποθήκες που τα μετατρέπουν σε μια εγκατάσταση κράτησης. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να τους καλύπτει, δεν υπάρχει καμία διαδικασία, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε κανένα δικαστήριο. Καταβλισμός θα πει ότι μπορεί να δουλέψει κάποιο εκεί. Όχι, δεν μπορεί κανείς να δουλέψει εκεί. Υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καθημερινή βάση σε αυτά τα μέρη. Για όσα μάλιστα ελέγχουν οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, τι να σα πω, δεν ξέρω και πόσα είναι όταν ε, έγινε στη Σαπορά τα πριν από 1,5 μήνα ε, μία ε, παρέμβαση, 15, μια επιχείρηση, 15.000 άτομα έφυγαν, μία ολόκληρη πόλη. τώρα τι συμβαίνει αυτό τι, σημαίνει, τι γίνεται στην, σε ολόκληρη τη Λιβύη, δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Πάντως ε, πάρα, ε, πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τη Σοβράτα και πήγαν στην Αλσούμ. Οπότε φαντάζεστε τι γίνεται στο σύνολο τη Λιβύη. Ε, σε κάποια τμήματα τη Λιβύη είναι μειωνοτικέ οι παραστρατιωτικέ οργανώσει. Είναι μειονοτικοί μάλλον οι, οι Έχουμε και πολλού ξένου. Δεν συμμετέχουν μόνο σε ανθρώπινο λαθρεμπόριο, αλλά προωθούν κάθε είδου λαθρεμπόριο εκτός Λιβύη λατρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών. Ε, αυτά είναι, είναι οι ίδιες παραστατικές οργανώσεις που προστατεύουν όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες και για να απαντήσω στο ερώτημά σας ε, ε, για τον εκπρόσωπο Αγγίλα, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές για το επιχειρηματικό ε, ε, ε, μοντέλο των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Ακολουθήστε απλώς το χρήμα, σαν να είναι τρομοκρατία, σαν να είναι ναρκωτικά, σαν να είναι οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Να δείτε από πού προέρχεται, ποιος αγοράζει πετρέλαιο που είναι συγκεκριμένο προϊόν προιον λαθρεμπορία, ε, ε, ε, ε, σκάφη με ευρωπαϊκές σημαίες που περνούν αυτό το λαθρέο πετρέλαιο κάθε μέρα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που εμπλέκονται στο ανθρώπινο, στο λαθρεμπόριο ανθρώπων. Λίγο περισσότερη αστυνομική δουλειά χρειάζεται, να συλλεχθούν οι πληροφορίες. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν απαγωγές, ζητούν λίτρα, ε, αυτό το αίτημα για λίτρα να κυκλοφορούν σε κοινωνικά μέσα δίνουν μάλιστα και λογαριασμούς στα σομαλικά, στα αραβικά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι ε, τραπεζικοί λογαριασμοί πού είναι αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί πολλοί από αυτούς είναι στην Ευρώπη. Κάποιοι άλλοι είναι στο ε, περσικό κόλπο. Ακολουθήστε το χρήμα και θα βρείτε τη λύση. Χρειαζόμαστε στενή αστυνομική συνεργασία σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Ξέρω ότι η, τα ευρωπαϊκά όργανα όλο και περισσότερο οργανώνεται για, να αξιοποιήσουν περισσότερο ε, τον ε, συντονισμό από την ενημέρωση, από τη Frontex, για παράδειγμα στην Ιταλία, αλλά για την ώρα μόνο Μωρισία υπάρχει. Δεν έχουμε ακούσει ένας λαθρέμπορος Μερικοί από αυτούς είναι και γνωστοί μάλιστα, έχουν αναφερθεί, έχουν κατονομαστεί από την ομάδα πυρογνωμόνων Κανένας από αυτούς ε, δεν έχουν ε, απαγόρευση ταξιδίου, ε, δεν έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί τους. Τι να σας πω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν είμαι αστυνομικός. Πάντως πρέπει να δοθεί προσοχή στις ροές χρημάτων. Αυτό θα προτείναμε στα κράτη να κάνουν όσον αφορά τον εθελοντικό επαναπατρισμό των μεταναστών. Ε, η επιστροφή είναι πάντοτε θελοντική. Αυτό ήταν το ερώτημα. Τις λίγες φορές που έχω πάει στη Λιβύη έχω δει ε, κόσμο να παρακαλά και να κλαίει για να γυρίσει στη χώρα του. Θέλει να γυρίσει στη χώρα του ή είναι πάρα πολύ απάνθρωπες οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης, ίσως ένα συνδυασμό και των δύο. Πάντως οι περισσότεροι θέλουν να πάνε σπίτι τους. Όμως πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό συστημάτων ε, για τη διάκριση ε, της κάθε κατάστασης και δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι έχουμε ένα μηχανισμό να, ε, που να εξασφαλίζει τέτοιες δικλείδες ασφαλείας για, για άτομα εκτός των 7 εθνικοτήτων που ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε πρόσβαση σε κάποια κέντρα κράτησης, ε, στο, ε, γύρω από την Βεγγάζη ε, που είναι υπό, την, ε, υπό τον έλεγχο του ε, απελευθερωτικού στρατού της Λιβύης όσον αφορά μιλήσατε για την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών, ναι, συμφωνώ, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας, πάντοτε θα ήθελα να αναφέρομαι στον Υπουργό Μπαζούμ, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών του Νίγηρα, είπε αν δεν υπάρχει ένα είδος ριζοσπατικοποίησης των νέων που βλέπει στην Αφρική, είναι ε, η ριζοσπαστικοποίηση ε, των, ε, του, του, της προσπάθειάς τους να βρουν ζωή αλλού. Αν τους πει κανείς ότι μπορούν να ζήσουν καλύτερα στη Λιβύη, να ζήσουν κάποια στιγμή καλύτερα αλλού, διασχίζοντας τη Μεσόγειο, δεν μπορείτε να τους αποτρέψετε. Εκτός εάν έχετε κάποιες καλύτερες συνθήκες υποδοχής στη χώρα που οδηγεί στη Λιβύη. Ε, ανεξαρτήτως λοιπόν του καθεστώτος πρέπει να αποτρέπουμε, που λαμβάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να τους αποτρέπουμε από το να φτάσουν στη Λιβύη, γιατί αν φτάσουν στη Λιβύη είναι πολύ αργά. Το ότι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε το σύστημα ασύλου, το σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης των, των, των χωρών που οδηγούν, ε, από, από τις οποίες περνούν για να πάνε στη Λιβύη, θα είναι χρήσιμο τουλάχιστον να μειώσουμε αυτό τον πειρασμό ε, των ανθρώπων να πάνε στη Λιβύη εθελοντικός επαναπατρισμός των προσφύγων. Λοιπόν, Κοιτάξτε, κάποιοι μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν. Η μεγάλη πλειοψηφία από το Ιράκ, από το Ιράκ, από την Παλαιστίνη, από την Ερυθρέα, από τη Σομαλία, περισσότεροι μπορεί να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ε, οι Σύριοι, οι Ιρακινοί, οι Παλαιστίνοι έχουν κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την καθημερινή του ζωή στη Λιβύη. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα προστασίας με την υποσαχά. Αφρική. Θα ήθελα να είμαι σαφή ω προ αυτό. Για αυτού ενδεχομένω να υπάρχει μια ανάγκη μετεγκατάσταση. Εμεί δίνουμε προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση για τους προερχόμενου από την υποσαχάρη Αφρική. Τι γίνεται με την αποβίβαση στα 12 σημεία αποβίβασης της ακτής της Λιβύης. Ε, συναντηθήκαμε με ομάδες του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε, ε, να δώσουμε τρόφιμα, να δώσουμε ε, ρουχισμό, να δώσουμε συμβουλές, ε, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, την, το λαθρεμπόριο ανθρώπων, ε, να μην πάρουν αυτούς τους ανθρώπους απλώς και να τους βάλουν στα κέντρα κράτησης και όταν επισκεφτόμαστε αυτά τα κέντρα ή μη, κάποιες μη, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που μπορούν να το κάνουν, μπορεί να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους διαφορετικά, χάνονται. Μερικές φορές μένουν εκεί, μερικές φορές φεύγουν, μερικές φορές πολλούνται, ε, γίνεται βουλεμπόριο δηλαδή. Αλλά έχουμε χάσει τα ίχνη τους μετά για την κατάσταση στο Βόρειο Νίγηρα Κοιτάξτε, ας μην ε, λέμε ψέματα σε σχέση με αυτά που μπορούμε να πετύχουν. Πράγματι υπάρχουν, ε, είναι επιτακτική πλέον η κατάσταση από, ανθρωπιστικές, ε, από ανθρωπιστικής απόψεως. Ας προσπαθήσουμε να σώσουμε όση πια ζωή μπορεί να σωθεί. Ας το κάνουμε αυτό, η υποστήριξή σας είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, να φύγουν οι πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές δυσκολίες ε, στη Λιβύη. Η κατάσταση στο Βόρειο Νίγηρα είναι προβληματική γιατί η κυβέρνηση του Νίγηρα δεν έχει μόνο υποδεχθεί πάνω από 200.000 ε, πρόσφυγες που έφυγαν ε, ξέφυγαν από τον Μπόκο Χαράμ ε, οι άλλες οργανώσεις από το κεντρικό Μάλι, ε, αλλά προσπαθούν ε, να βοηθήσουν τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια παράκαμψη πλέον έξω από τον ήγυρα που πηγαίνουν στη Λιβύη, με, άλλο, με άλλη διαδρομή. Ε, πολλοί άνθρωποι ε, έχουν γίνει λαθρέμποροι και μετά η κυβέρνηση τους είπε ότι α, δεν, μπορείτε πια, δεν μπορείτε πια να είστε λαθρέμποροι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια άλλη οικονομία, μια εναλλακτική οικονομία. Οι τοπικές αρχές καλούν όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, που συμμετείχαν στο εμπόριο αυτό να εμφανιστούν, υποσχόμενοι όχι αμνηστία, αλλά τέλος πάντων μη δίωξη. 5.000 άτομα ε, μάλιστα εμφανίστηκαν και είπαν ε, ότι ε, όντως ε, είχαν συμμετάσχει και προσπάθησαν κάπως να τους βοηθήσουν να φύγουν από αυτήν την κατάσταση να μετατρέψουν τέλος πάντων αυτή την παραοικονομία σε οικονομία. γιατί όντως ε, χάνονται και πάρα πολλά εισοδήματα στο Βόρειο Νίγηρα μέσω αυτής της, παραοικονομία. της παραοικονομίας. Ε, θα θυμάστε την εικόνα του Αιλάν ε, στην ακτή ενός νησιού στην Ελλάδα τόσα πολλά, τόσες πολλές αναφορές στα κοινωνικά μέσα ε, υπάρχουν κάθε μέρα ε, για το τι γίνεται στην Αφρική. Από απόψεις υποστήριξης είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι απλώς να υποστηρίξουν ε, την ακτοφυλακή της Λιβύης αλλά και άλλους θεσμούς ε, κατά της διαφθοράς, τους τον εισαγγελέα, όλους όσους ε, προσπαθούν να ε, βοηθήσουν τη Λιβύη να ε, σεβαστεί τις δεσμεύσεις της. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όλους όσους προσπαθούν να αλλάξουν τη χώρα αυτή. Μίλησα ήδη για την κατάρριψη του επιχειρηματικού πλάνου των λαθρεμπόρων. Ο Νίγηρας ε, δέχεται τους πρόσφυγες που έρχονται στον Νίγηρα αλλά και αυτούς που θα εκενωθούν από τη Λυφή, ε, με διάφορες πτήσεις από αύριο εκτός ε, από την εκ νέου ένταξη των δικών τους υπηκών, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών θα βρούμε μία λύση εξόδου σε άλλες χώρες στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες του κόσμου. Όσον αφορά τη δημοσίευση των αριθμιστικών στοιχείων για όσους πηγαίνουν ε, στη Λιβύη, είναι στατιστικές της Eurostat. Τις χρησιμοποιούμε. Προφανώς αν είχαμε περισσότερο νόμιμες εναλλακτικέ ε, όσον αφορά την καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις περισσότερες, σε περισσότερες χώρες διέλευσης, ε, πολλοί δεν θα αισθάνονταν υποχρεωμένοι να προχωρήσουν. Υπάρχει μια διαφορά δέσμευσης μεταξύ ε, Σουδάν και η Αιθιοπία. Σε Αιθιοπία έχουμε τώρα μια πολιτική εκτός των καταβλισμών, το δικαίωμα εργασία των προσφύγων, οπότε βλέπουμε πρόοδο, βλέπουμε λιγότερους Ερυθρέου να φεύγουν από την Αιθιοπία για να πάνε μέσα από τα δάση στη Λιβύη, αλλά 80% των Ερυθρέων φτάνουν στο Σουδάν και συνεχίζουν προ Αίγυπτο και Λιβύη. Οπότε βλέπουμε ε, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν υπηρεσίες ε, τοπικά και αυτό μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά όσον αφορά την ε, σταθερότητα των προσφύγων, την αξιοπρέπειά τους και να τους δίνουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα που πρώτα ζήτησαν άσυλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ε, οι απαντήσεις σας. Ο κύριος Καπρίτσι, η Βικυρία Μπιλαρόσα από την ΕΚΟ. Εσείς παρακαλώ. Μόνο 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα θέλω να υπογραμμίσω ότι εμείς συνεργαζόμαστε με, το Διεθνή, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ε, για πάνω από δύο χρόνια για το θέμα αυτό και το θέμα της προσέγγισης είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ και πολύ καιρό αυτά που είπε το CNN. Το θέμα είναι ότι όταν κανείς ε, τα λέει αυτά στα κράτη-μέλη ανεξάρτητα από ε, την εντύπωση που προκαλείται στην κοινή γνώμη το ότι η Ευρώπη στέλνει ανθρώπου πίσω, κατ' ουσίαν κανεί δεν ασχολείται με την ανθρωπιστική διάσταση. Επιστρέφουν άνθρωποι σε εμφύλιο πόλεμο. Εμείς ε, προσπαθούμε λοιπόν να το προβάλλουμε αυτό, ε, την υποστήριξη των κρατών μελών. Βέβαια το CNN ήταν καθοριστικό και καταλητικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το CNN το βλέπουν παντού και κατά δεύτερον, ακόμα και δεν είναι κάτι καινούριο, είναι η πρώτη φορά που μετά το CNN είχαμε την πρόταση από τη Ρουάντα να δεχτούν 30.000 ανθρώπους. Αν μία χώρα πει ότι αυτό είναι ανθρωπιστική καταστροφή, αυτή είναι δουλεία, αυτή εκεί είναι αδελφοί μας, εγώ προσφέρομαι να αναλάβω μερικούς, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η αρχή, μετακολουθούν και άλλοι και με την δήλωση που είναι πολύ γενική και ασαφής, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια κίνηση από όλες τις αφρικανικές χώρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, και η αρμοστία και ο Διεθνής Οργανισμός αρχίζουν να δραστηριοποιούνται σε αυτό που είχαμε ήδη ξεκινήσει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει κανείς την υποστήριξη των υποσαχάριων χωρών ε, μόνο για τις ε, οικειοθελείς επιστροφές. Να υπάρχει δηλαδή μία προθυμία και ένα συντονισμός. Ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, ε, συν η δήλωση της Καγκάμε, αυτά μας έφεραν σε αυτήν την κοινή δήλωση. Τώρα, πώς, ποιο θα είναι το περιεχόμενο της δήλωσης ακριβώς, κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Έχουν λάβει χώρα κάποιες τεχνικές συζητήσεις. Είναι όμως πολύ σημαντικό το ότι να ξέρουμε ο μηχανισμός δεν είναι τέλειος, αλλά από πλευράς αριθμού υπάρχουν, υπάρχει, υπάρχουν αρκετοί και επειδή δεν μπορούμε να πούμε στα κέντρα, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η δήλωση. Άρα δηλαδή να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το δυναμισμό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Υπάρχει πάντως ε, κάποια ευκαιρία. Τώρα για την κατάσταση στη Λιβύη, ε, αυτή είναι πολύ ευμετάβλητη. Ε, κάποιοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει business ε, με την κυβέρνηση της Λιβύης. Οι άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να διπραγματευτούμε είναι πάρα πολύ λίγοι. Πράγματι υπάρχει αυτό το στοιχείο της συνευτικής διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών, αυτή τρέχει, αυτή η διαδικασία και όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, όταν η Λιβύη ήταν σταθερή, μιλάμε τότε για δύο εκατομμύρια ανθρώπους, ε, μη Λιβύους που ζούσαν και εργαζόντουσαν ε, στη Λιβύη. Αυτή τώρα σήμερα είναι 750.000. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, το πού βρίσκονται τα χρήματα, πού βρίσκονται οι λαθροδιακινητές. Αυτά είναι καθοριστική σημασία. Εμείς ε, έχουμε δουλέψει σε αυτό η ε, επιχείρηση Σοφία δεν είναι για να επιστρέψουν οι άνθρωποι, να τους διώξουν, αλλά πρόκειται για την ε, συλλογή ε, πληροφοριών. Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, η Σοφία, το, ο μηχανισμός αυτός να έρθει σε επαφή με τη Europol, τη Eurojust και πολλά άλλα. Όμως όλα αυτά είναι ένα στοιχείο για να διαταραχθεί το επιχειρηματικό μοντέλο. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι λαθροδιακινητές με την έννοια ότι ήταν ανέκαθεν εγκληματίε. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι κανονικοί άνθρωποι, είχαν παλαιότερα κάποια δουλειά ασχολιόντουσαν με το ε, κτήμα τους. Σε αυτήν όμως την κατάσταση, όσο έχει διαμορφωθεί στη Λιβύη, πάνω από 500.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι Λιβύοι για να ζήσουν μόνο λένε εντάξει παλαιότερα ήμουν βοσκός αλλά αν μπορώ και εγώ να βγάλω κάποια χρήματα ε, με τη μεταφορά ανθρώπων ασχολούνται και αυτοί με τη δουλειά χωρίς να ασχολιόντουσαν στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, ε, σταθεροποίηση της Λιβύης και αναδιάρθρωση το, της τοπικής κοινωνίας όπου επαναλαμβάνω και πάλι εκεί ζούσαν πολλοί μη Λίβοι, αυτό είναι καθοριστική σημασία. Αυτό που κάνουμε, ε, η αποβίβαση, η ταυτοποίηση, αυτά είναι φιάλτης αλλά είναι η μόνη δυνατότητα για να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από τη σκλαβιά. Ας ε, επικρίνουμε, ας ασκούμε κριτική, καλό, σωστό αυτό, αλλά και πρέπει παράλληλα να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να βρεθεί ε, κάποια λύση. Άρα, σύν συν οι δηλώσεις του Καγκάμε, αυτό είναι μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Κυρία Βιλαρόσα, από τη Γενική Διεύθυνση δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Μα πιέζει ο χρόνο. Ούτω ή άλλω, τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν δύο λεπτά το πολύ χρόνο αγόρευση στην Ολομέλεια. Δεν το κάνουμε για εσά, ούτε και εμεί έχουμε πολύ. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρω. Όπως γνωρίζετε, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να βασίζεται ε, σε συγκεκριμένο καθεστώς, ε, βασίζεται σε αρχές. Και να υπενθυμίσει αυτό που είπε και ο κύριος Κοστέλ στην αρχή. Έχουμε μισό εκατομμύριο Λιβύους οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι άτομα τα οποία χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και φυσικά υπάρχει η κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων. η κατάσταση επιδεινώνεται. Έχουμε γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους που έχουν χάσει ε, τη στέγη τους και τα υπάρχοντά τους, εσωτερικώς εκτοπισμένους που είναι υποχρεωμένοι να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους ε, για να επιβιώσουν, πολίτες οι οποίοι βρίσκονται μέσω ε, αντίπαλων ομάδων ή στα χέρια του Ισλαμικού κράτους ή άλλων τρομοκρατικών ομάδων. Έχουμε ασθενείς που τους έχει επηρεάσει κατάρρευση του συστήματος υγείας και βεβαίως και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ε, να τύχουν φροντίδας. Γι' αυτό ακριβώς ε, και το ανθρωπιστικό μέσο ΕΚΟ ε, επικεντρώνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, σε στενό συντονισμό και σε συμπληρωματικότητα των άλλων ευρωπαϊκών μέσων, κυρίως εκείνων που στοχεύουν περισσότερο στην μεταναστευτική κρίση και το 2018 θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε κυρίως στον τομέα της υγείας όπως ανέφερα. Πρόκειται για έναν από τους τομείς που έχουν πληγεί κυρίως από την κρίση στη Λιβύη και θα ήθελα να σας δώσω κάποια λίγα στοιχεία. Λιγότερο από το 20% των εγκαταστάσεων υγείας λειτουργούν σε κάποιες γειτονιές. Ε, Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι δεν υπάρχει τακτική πρόσβαση σε φάρμακα, ε, μόνο ε, κάποιες κλινικές λειτουργούν πλήρως και μόνο 40% των ε, βασικών παροχών για παιδιά και κλινικές λειτουργούν. Από τη Γενική Διεύθυνση Νίερο, ο κύριος Λόρη. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι γνωρίζω ότι ο χρόνος τρέχει. Να σας πω απλώς ότι οι δραματικές συνθήκες ε, ε, στις οποίες ζουν οι μετανάστες ε, στη Λιβύη και που μας ανέφερε ο κύριος Κοστέλ εδώ σήμερα δείχνουν ότι πρέπει κατεπηγόντως να δράσουμε στη χώρα αυτή και υποστηρίζουν πλήρως την στήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αξιοθαύμαστες προσπάθειες οργανώσεων όπως ε, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Υπατή Αρμοστία για, την πρόσθε, ε, για τους πρόσφυγες και κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσει που παρά τι επονίδιστε συνθήκε ε, στη χώρα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται. Να σα πω ότι το καταπιστευματικό Ταμείο Κατεπίγουσα Βοήθεια για την Αφρική και κυρίω για τη Βόρεια Αφρική θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και κάποιε άλλε οργανώσει το 2018 και τη στιγμή που σα μιλάω τώρα, η Επιχειρησιακή Επιτροπή του Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική αποφάσισε την εκταμείευση ενό σημαντικού ε, ποσού για την καταπολέμηση τη της ε, λαθροδιακίνησης ε, ε, μέσω του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές και να πω για τους συναδέλφους ότι ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία σοκάρουν. Ε, πιστεύω και ότι και οι χώρες μας μπορούν να κάνουν περισσότερα. Ερωτήσεις για το ποιο δίνει άδειε στα σκάφη αυτά για να δραστηριοποιούνται. Πού είναι οι λογαριασμοί τραπέζι όλων αυτών των ανθρώπων. Ε, πολύ ωραία και καλά λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο το άλλο. Χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των χωρών όμως για να δράσουμε. Έχουμε ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Ε, οι συνάδελφοι όμως ψηφίζουν στις πολιτικές ομάδες ε, τους ε, για την επόμενη εβδομάδα. Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε συνέχεια στο Αμπιτζάν, να θέσουμε αυτές τις ερωτήσεις και να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά, διότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κωστέλ, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στο σημείο 10, στα διάφορα. Κανείς δεν έθεσε καμία ερώτηση για το σημείο 11 και η επόμενη συνάντηση είναι στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η τελευταία επίσημη συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα. Έχουμε τη συνεδρίαση για το βραβείο Ζαχάροφ την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να σας δω, ε, αλλά ε, αν δεν σας δω, καλές γιορτές. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς πρόεδρος.